Okay, dear colleagues, let's start uh, with point Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε με το σημείο 9 της ατζέντα. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των τεχνολογικών προτύπων, η πληροφορία τη Εταιρεία των Διεθνών Προτύπων Χρηματικών Αναφορά τη Ευρωπαϊκή Ελληνική Ομάδα για τα θέματα χρηματοοικονομική αναφορά. Τέσσερι γραμμέ ε, είναι ο τίτλο και αυτό αποτυπώνει την περιπλοκότητα του ζητήματος. Δεν θα σας διαβάσω όλα. Θα δώσω πάρα αυτά το λόγο στον εισηγητή μας, ο οποίος είναι ο κύριος Στόλογιαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η επένδυση είναι βασικός ε, Κινητήρα τη ανάπτυξη και των θέσεων απασχόληση και τα διεθνή λογιστικά λοιπόν πρότυπα είναι απαραίτητα για την καλή ποιότητα και την αξιοπιστία των σχετικών πληροφοριών. Σήμερα λοιπόν που εφαρμόζονται το 2005 τα διεθνή λογιστικά πρότυπα ε, και χρησιμοποιούνται 160 χώρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά λοιπόν τα πρότυπα αυτά για την καλή λειτουργία των κεφαλαίων και θεωρούνται λοιπόν δημόσιο αγαθό υπό την έννοια αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να είναι διαφανή, ανεξάρτητα και να υπόκειται στο δημόσιο έλεγχο. Η οικονομική κρίση έθεσε το θέμα των διεθνών λογιστικών προτύπων και του αντίκτυπου στις τράπεζες στην ημερήσια διάταξη του G20 αλλά και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων μεταξύ άλλων και του Κοινοβουλίου. Η ΕΚΟΝ δημιουργεί σε μια μόνιμη ομάδα εργασίας για το θέμα. Και έθεσε το θέμα της ποιότητας και της ε, διαχείρισης των διεθνών λογιστικών προτύπων καθώς και τη ΕΦΡΑΓ για την περίοδο 2014-2020. Η έκθεση αυτή φέρει το όνομά μου. Αλλά για να είμαι δίκαιος θα πρέπει να πω ότι μόνο χάρη στο σεμινάριο και στις ακριάσεις ε, μπορέσαμε να βγάλουμε κάποια άκρη. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Σας ευχαριστώ και για τη συμμετοχή σας και για την συμβολή σας. Για την έκθεση. Τι θέλουμε να πετύχουμε με την έκθεση σε ό,τι αφορά την ποιότητα των προτύπων. Κοινή κατανόηση του κριτηρίου δημοσίου αγαθό τα πρότυπα αυτά δεν θα πρέπει να διακυβεύουν ούτε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε να αποτρέπουν και την ανάπτυξη. Για να υποστηρίξουμε την ε, πρόταση του ICRB σε ό,τι αφορά την αρχή της πρόληψης και για να υπάρξει και μεγαλύτερη υποστήριξη προς τις αρχές αυτές που συνάντουν με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ICB και η ΕΦΡΑΓ, η Πολιτική Ομάδα για τα Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Θα πρέπει να λάβουν υπόψη ε, τις αντίκτυπο των προτύπων αυτών και θα πρέπει να γίνουν απολύτω κατανοητά τα πρότυπα αυτά. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή, ότι λόγω ακριβώ και χάρη τη ε, συμβολή ε, του Κοινοβουλίου, η ICB και η ΕΦΡΑΚ επιδεικνύουν πλέον ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά την ανάλυση αντικτύπου. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχουν σε μια πρώιμη φάση κατάρτισης των ε, διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς και ο διάλογος μεταξύ ISCB και τη συμβουλευτική ομάδα θα πρέπει να συνεχίσει παρά την ε, διαδικασία σύγκληση. Τώρα, για διακυβέρνηση του IFRS ε, και τη EFRAG. Θα πρέπει να κοιτάξουμε θέματα εσωτερική οργάνωση μέχρι και τη συζήτηση δημοσίου συμφέροντος, τα οποία θα πρέπει να δοθούν προ το Ίδρυμα IFRS. Η χρήση των ε, διεθνών προτύπων και η μόνιμη χρηματοοικονομική συνεισφορά θα πρέπει να είναι όρη για τα σώματα εποπτείας και παρακολούθησης του Ιδρύματος IFRS και του ICB. Και η έκθεση μάλιστα το έχει συμπεριλάβει διάφορες απαραίτητες συστάσεις. Και γι' αυτό λοιπόν για την ΕΦΡΑΓΑ για την περίοδο 2017 μέχρι 2020 ε, θα πρέπει να εξετάσουμε τι θα γίνει, γιατί όταν εγκρίνουμε ένα πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Κοινοβούλιο, η ε, η χρηματοδότηση ήταν μόνο για το 2014 μέχρι το 2016. Τώρα για το, τα καινούργια διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφορά. Ε, ήταν θετική η γνωμοδότηση της ΕΦΡΑΚ σχετικά και περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για πράξεις κατά εξουδιοδότηση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Και εκ παραλλήλου λάβαμε ασφαλώ και δημόσια θετικές ε, εντυπώσεις από την ΕΚΤ, από άλλα θεσμικά όργανα για τα διεθνή πρότυπα. Το IFRS 4 για τις ε, ασφαλιστικές είναι που εξέλιξη και η ΕΚΤ πρότεινε για την εφαρμογή των διεθνών προτύπων αναφοράς Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο εισήγητη. Θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις των πολιτικών ομάδων. Εξ ονόματος ε, της κυρίας Πέρες, η κυρία Γκίλ. Δυστυχώς η περδόνσο δεν μπορεί να είναι παρούσα, όπως είπατε είναι η σκιώδης εισηγήτρια για τα θέματα αυτά, ζητά συγγνώμη. Θέλει να ευχαριστήσει τον κύριο Στόλογιαν για την πρότασή του. Θεωρεί ότι πράγματι αντικατοπτρίζει η πρόταση τα θέματα που έθεσαν τα μέλη της ΕΚΟΝ στα πλαίσια της ομάδας εργασίας IFRS. Έγιναν χρήσιμες συζητήσεις και με τους εκπροσώπους της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας και με τους εκπροσώπους της Επιτροπής και με τους εκπροσώπους της ΕΦΡΑΓ για το IFRS 9. Υπήρξαν λοιπόν αρκετά θετικά στοιχεία στην πρόταση. Η αντίληψη η οποία διέπει την έκθεση ότι δηλαδή τα κριτήρια Μάισταντ και η δημοσιονομική σταθερότητα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια των διαδικασιών έγκρισης. Τα κριτήρια αυτά είναι στην καρδιά της προστιθέμενης αξίας σε σχέση με τα λογιστικά πρότυπα της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής. Ταυτόχρονα η κυρία Μπερές υποστηρίζει ότι έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος σχετικά με την μεταρρύθμιση EFRAG και ότι τώρα θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να περάσουμε στην εφαρμογή αυτών που έχουν προταθεί πριν υπάρξει διεύρυνση του κοινοτικού προγράμματος για το EFRAG για την περίοδο 2020, 2017 συγγνώμη, 2020. Ταυτόχρονα συμφωνεί με τις ανησυχίες για ένα νέο πρόεδρο για την ΕΦΡΑΓ. Η διαδικασία για την πρόσληψη του νέου αυτού προέδρου είναι ιδιαίτερο αργή και αυτό θα βλάψει την ποιότητα της λειτουργίας της ΕΦΡΑΓ. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ακουστεί επιτέλους η ευρωπαϊκή φωνή. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές τις οποίες προτείνουμε για την ε, συγκεκριμένη πρόταση στο Υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την διακυβέρνηση του IFRS και του IASB όπως επίσης και τα λεγόμενα και για το Συμβούλιο Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος, το οποίο θα λέμε από εδώ και πέρα PIOB. Ε, όλα αυτά και ιδιαίτερα το τελευταίο είναι βασικά συστατικά για να μην υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων. Ε, σχετικά τώρα με το IFRS 9 ε, αναφέρεται σε ένα εδάφιο, θα ήθελα να υπάρξει μεγαλύτερη αναφορά για το νέο αυτό κανόνα των χρηματοοικονομικών μέσων υπογραμμίζει την σημασία που υπάρχει για το IFRS 9 να εξυπηρετήσει την μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Θέλω να υπογραμμίσω επίσης ότι αυτά τα λογιστικά πρότυπα θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρότερα υπόψη θέματα φορολογίας και πιθανότητες φορολογικής απάτης. Τέτοιες πλευρές αγνοούνται μερικές φορές Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην παρούσα συγκυρία. Να προσθέσω και εγώ ως γκυλ ένα πρόσημο. Θα υποστηρίξω πλήρως την ανάγκη μεγαλύτερης σύγκρισης ε, και ανάγκη γενικότερα ευρύτερης χρήσης ε, των εκθέσεων και των ανακοινώσεων σχετικά με την υγεία μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. Για να γίνει αυτό βέβαια ε, πρέπει να υπάρξει μια κοινή γλώσσα και αυτό μπορεί να γίνει και σε σχέση ε, με τα δελτία ε, τα οποία εκδίδονται για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σουίνμπορν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδεις για τη δουλειά που έκαναν μέχρι τώρα και να μεταφέρω τις απόψεις του Σάιντ Καμάλ που ζητά συγγνώμη γιατί είναι απόν σήμερα. Ευχαριστεί τον εισηγητή για μια πολύ προσεκτική και ισόρροπη έκθεση. Λέγει ότι το θέμα έχει συζητηθεί αρκετά μέχρι τώρα. Η χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε ότι οι μεταρρυθμίσεις απαιτούνται πλέον ε, και σήμερα ε, συζητάμε ένα βελτιωμένο σύστημα λογιστικών προτύπων. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν πάρα πολλές δυσκολίες μέχρι το τέλος του προηγούμενου χρόνου. Υπήρξαν αμφιβολίες όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα των λογιστικών προτύπων, των λογιστικών διαδικασιών, ε, θα πρέπει να υπάρξει εξέταση του ρόλου που έχει παίξει το IAS 39 ε, και που οδήγησε στην ε, πτώχευση ουσιαστικά αυτού του οργανισμού. Νομίζω ότι όλοι βέβαια ασφαλιστές, τραπεζίτες, λογιστές έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το τι πρέπει να περιλαμβάνουν τα δελτία και οι απολογισμοί των επιχειρήσεων και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια σύγκληση εδώ. Ε, ένα IFRS δεν θα πρέπει να είναι αντίθετο ε, με τις βασικές αρχές της λειτουργίας της αγοράς. Αν κάτι τέτοιο ισχύει τότε δεν μπορεί να γίνει φυσικά δεκτό. Η έννοια του true and fair view είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στους απολογισμούς των επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι αριθμοί δεν θα πρέπει να είναι ούτε υπερβολικοί ούτε και κρυμμένοι. Αυτό νομίζω ότι ε, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και στα πλαίσια της, ε, των προβλεπομένων της οδηγίας της διατήρησης κεφαλαίων. Αν υπάρξουν λάθη θα μπορούσαμε σε μερίσματα τα οποία θα μπορούσαν να πληρωθούν ως μιέδη. Ο Δόκτωρ Καμάλ λοιπόν πιστεύει ότι απαιτείται μια πιο λεπτομερής περιγραφή της αρχής του True and Fair View. Ε, θα ήθελα να πω ότι η αξιολόγηση για το IFRS πρέπει να συνεχιστεί. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση εκ νέου για το IFRS 4 σχετικά με τις πιθανές καθυστερήσεις της εφαρμογής του συγκεκριμένου κανονισμού για ασφαλιστικές μονάδες στο εσωτερικό των πιστοτικών ιδρυμάτων. Ευχαριστώ. I guess from Alde is... Ο κύριος Γιάτσεκ από την Άλντε θα είναι πάλι φαντάζομαι. Ναι, ευχαριστώ. Σωστά, έχετε δίκιο. Εξ ονόματος ε, της Κόρα. Ε, Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τα όσα μας παρουσίασε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα οποία να είναι συγκρίσιμα και ομοιόμορφα και έτσι να αυξηθεί περαιτέρω η διαφάνεια. Δεύτερη... Δεύτερον, τα διεθνή πρότυπα είναι σημαντικά για το εμπόριο, τον ανταγωνισμό, αλλά και για την άρση των επενδυτικών φραγμών. Πιο συγκεκριμένα, η ε, ΚΟΡΑ υποστηρίζει την ε, σημασία της ε, σωστής ανάλυσης αντικτύπου, της καταπολέμησης των, της περιπλοκότητας, αλλά και έναν επικοδομητικό διάλογο ανάμεσα στην ISB και στην ομόλογό της, τον ΙΠΑ. Ε, είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να βρούμε σωστή ισορροπία ανάμεσα στην περιπλοκότητα και την απλότητα. Οι προδιαγραφές θα πρέπει να είναι, τα πρότυπα θα πρέπει να είναι καθολικά και διαφανή και να αντικατοπτρίζουν την οικονομική πραγματικότητα. Ε, προσβλέπουμε στην περαιτέρω συμβολή μας ε, τι επόμενες εβδομάδες αυτή την εργασία και θα συνεργαστώ με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους κοιόδης. Ευχαριστώ, Ντεμάση για την Γκούέ. Καταρχά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης. Έχω να διατυπώσω τρία σχόλια σε αυτή τη φάση, ότι η ISP και η Έφρακος ε, είναι ιδιωτικές ε, ε, οι οποίε υποτίθεται θεσπίζουν ε, διεθνή πρότυπα προ το δημόσιο συμφέρον. Όμω ξέρουμε από την κρίση ότι οι μέθοδοι αξιολόγηση ε, μετράνε όχι μόνο για την μέτρηση της πραγματικότητας, αλλά και έχουν μακροοικονομικές ε, σοβαρές συνέπειες και γι' αυτό θέλουμε να δούμε ποιες άλλες ομάδες ενδιαφέρονται για αυτά τα πρότυπα για να αποφύγουμε πιθανά πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και θα θέλαμε αυτά τα όργανα να μετατραπούν σε δημόσιους οργανισμούς ώστε να υπάρχουν υπάρχουν και... Α, και αυτό θέλουμε αυτό να αντικατοπτρίζεται στο εκτιμώντα σε κάπα. Για την περιπλοκότητα και το άρθρο 5 συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε απλούστερες προδιαγραφές και πρότυπα, αλλά μας ανησυχεί και η οικονομική, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Πιστεύουμε πως έχουμε πιο περίπλοκια πρότυπα αυτή τη στιγμή, αλλά ωστόσο δεν αντιμετωπίζονται θέματα όπως η αναγνώριση τη ζημιά και ε, οι δυνητικές ε, αρνητικές επιπτώσεις ε, Επίση, είμαστε κάπως διστακτικοί όσον αφορά τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 8. Μπορεί να είναι χρήσιμα, αλλά σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο θα πρέπει πολύ προσεκτικά να σκεφτούμε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις και δεν ξέρουμε κατά πόσο ε, λαμβάνονται όλα υπόψη σε οποιοδήποτε πρότυπο, ώστε να υπάρχει, θέλουμε να υπάρχει πάντοτε επαρκής εκπροσώπηση σε αυτά τα όργανα. Ευχαριστώ, Σφέν Γίγκολτ, εξ ονόματος των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ, κύριε Στόλογιαν, για την έκθεσή σας. Έχετε λάβει υπόψη τις συζητήσεις που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και θέλω να αναφέρω κάποια σημεία όπου θα πρέπει να βασιστούμε στα όσα έχουμε ήδη πει και να προσθέσουμε. Ε, καταρχάς, όντως η παγκοσμιοποίηση και οι παγκόσμιες κεφαλαγορές θα μπορούσαν να ωφεληθούν, όπως είπε και η Νίνα Γκίλ, από πιο ομοιόμορφους και συγκρίσιμους κανόνες. Απ' την άλλη, αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι κανόνες θεσπίζονται σε ένα διεθνές επίπεδο ε, όμως ο τρόπος με τον οποίο θεσπίζονται θα πρέπει να αντιστοιχεί με τις αρχές τις οποίες μόλις ψηφίσαμε στο πλαίσιο της έκθεσης Γκουλάρ, δηλαδή δημοκρατική νομιμότητα, διαφάνεια, κεραιότητα και λογοδοσία. και η ISB παρά τις πρώτες κινήσεις που βοσίζονται στις συστάσεις μάισταντ, δεν πληρεί όλα αυτά τα κριτήρια. Ο κ. Στόλογιαν στην έκθεσή του επίσης αναφέρει, αναφέρεται σε κάποια από τα προβλήματα και πιστεύω θα πρέπει πλήρως να εφαρμόσουμε τα πρότυπα από των οποίων μόλις ψηφίσαμε στην ΕΚΟΝ στο πλαίσιο της έκθεσης Γκουλάρ για το IFRS και το ISB και για το EFRAG, το οποίο επίσης, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όντως ισχύει η δημοκρατική νομιμότητα, η διαφάνεια, η κυριότητα και η λογοδοσία. Στηρίζουμε και θα θέλαμε να ενισχύσουμε αυτό το τομέα της ε, μελέτης αντικτύπου, Βεβαίως και με τα κριτήρια έγκρισης που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε τις δυνατότητες, για παράδειγμα μακροοικονομική ανάλυση ως προς αυτό το σημείο. Πέραν τούτου είναι σημαντικό η Ευρώπη να μιλά με δυνατή φωνή όταν πρόκειται για παγκόσμιες διαδικασίες θέσπισης προτύπων. Και το βασικό θέμα με την λογοδοσία είναι ότι αυτή τη στιγμή το όργανο εποπτείας που έχει φτιαχτεί δεν συμφωνεί, τα, έργανα μάλλον εποπτείας δεν συμφωνούν αν θέλουν να είναι εποπτικό συμβούλιο ή όχι. Ένα εποπτικό συμβούλιο που δεν συμφωνεί εάν θέλει να λαμβάνει ουσιαστικέ αποφάσει. δεν έχει να κάνει μόνο με θέματα δημοσίου συμφέροντος, αλλά με το κατά πόσο το εποπτικό αυτό συμβούλιο θέλει να είναι ο θεματοφύλακας του θεσμού και εφόσον μπορεί να αποφασίσει μόνο με συνένεση, αυτή τη στιγμή επικρατεί ε, μια, ε, ένα, μια, ένα πάγωμα της κατάστασης και στην ουσία το ISB ε, ελέγχει τον εαυτό του. Και αυτό είναι αμφίβολο και από ευρωπαϊκή προοπτική, γιατί έχουμε βάλει πολλά χρήματα εκεί. Νομίζω λοιπόν πως είναι πολύ σημαντικό ο ρόλος του Εποπτικού Συμβουλίου να αποσαφινιστεί και να παρέχει όντως την καθοδήγηση αυτό το όργανο και εφόσον δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί θα πρέπει να τεθούν θέματα νομιμότητος. Έπειτα, σύσταση, συστάσεις μάλιστα για το δημόσιο συμφέρον. Συμπεριλαμβανομένες της ανάγκης συμβολής στην οικονομική σταθερότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να ληφθεί πλήρως υπόψη στη διάρκεια της διαδικασία έγκριση και το σχέδιο έκθεση αυτό το τονίζει. Είναι όμως εξίσου σημαντικό να ενσωματώνονται όλα αυτά στον τρόπο με τον οποίο ε, ε, η ISB ε, συστήνει τις, τα πρότυπά τη και κατά πόσο θα είναι δεσμευτικά τα κριτήρια έγκριση. Είναι δύσκολο τα ισχύοντα πρότυπα να αναφερθούν σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια, γιατί αν αλλάξει κανείς τα κριτήρια είναι κάτι, αλλά η λογική συνέπεια αυτού είναι βεβαίω ότι τα διάφορα πρότυπα θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτά τα κριτήρια. Αυτό που είναι σημαντικό όσον αφορά την ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι ότι ο βασικός γνώμονας για μας εδώ όταν κάναμε τις ε, οικονομικές ε, μεταρρυθμίσεις ήταν η έκθεση Ντελαροζιέ όπου οι περισσότερες συστάσεις καταφέραμε να τις λάβουμε υπόψη. Αλλά η έκθεση Δελαροζιέ είναι γεμάτη με συστάσεις για τα λογιστικά πρότυπα και τον κίνδυνο της προκυκλικότητας και αυτό το κομμάτι της ατζέντα μεταρρύθμισης δεν έχει ολοκληρωθεί. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την έκθεση θα πρέπει να, να σημειώσουμε την έκθεση Ντελαροζιέ και να εξετάσουμε μέχρι ποιο σημείου η ISB έχει όντω ε, υλοποιήσει αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Τέλο, όσον αφορά τα ίδια τα πρότυπα και την ουσία του και όσο αυτά δεν λαμβάνουν υπόψη την αληθινή και δίκαιη οικονομική σταθερότητα, θα είναι αμφίβολη έκκληση αν δεν τα επεκτείνουμε για τις μικρομεσαίες ή τις μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις. Αυτό θα πρέπει να γίνει μόνο όταν τα πρότυπα θα είναι σωστά και όταν, για παράδειγμα, οι κανόνες market to market για ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα κυριαρχούν, αυτό θα πρέπει να ξεπερνούν την εντολή που ήδη έχουν. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η FTD δεν πλάκω κανέναν. Μπάρμπαρα Κάπρα, ναι. möchte. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ ισορροπημένη αυτή έκθεση και συμφωνώ με την εκτίμηση ότι είναι σημαντικό να κοιτάξουμε τα θέματα αυτά στην αξιολόγηση μας, στην αξιολόγησή μας και ότι στην e ISB τα πράγματα πάνε καλά, στην ISB. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα είναι σημαντικά για την ανταγωνιστικότητα και για τα κεφάλαια και για τις επενδύσεις στις επιχειρήσεις και γι' αυτό θεωρούμε ότι Καλωσορίζουμε αυτή την ε, πλαισίωση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο γιατί πρόκειται για ένα σημαντικό τμήμα του πλαισίου ρύθμιση, στο πλαίσιο των ε, υπηρεσιών των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της ΕΣΜΑ. Κάποια σημεία τα οποία μου φαίνονται ότι είναι σημαντικά σε ό,τι αφορά το EFRS και τα οποία τα έφερε και ο συγητής είναι πολύ περίπλοκη η υποχρέωση αναφορών Χαίρομαι επίσης ότι για το ότι υπάρχει έκκληση να αναπτυχθούν ξεχωριστά πρότυπα για τις μικρομεσαίες και τέλος θέματα συνοχή και ομοιογενοποίησης. Καταρχά. σημαντικό είναι το συμφέρον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι σημαντικό το έργο της ΕΦΡΑΓ και θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε και ενδεχομένω θα υπάρχουν και περαιτέρω θα πρέπει να υπάρξουν και περαιτέρω μέτρα υποστήριξη τη ΕΦΡΑΓ θα συμμετάσχει φαντάζομαι και το EFRS, ε, η ομάδα του Κοινοβουλίου. Και τέλος, ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, ε, για παράδειγμα με τις ΕΙΠΑ, που είναι στο τέλος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, είναι σκόπιμο τα πρότυπα αυτά να αναρμονιστούν σε παγκοσμίο επίπεδο και προς την κατεύθυνση αυτή θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να ζητάει το, λόγο, το λόγο στην διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ. Άρα, να δώσουμε το λόγο πάλι στην, πάλι στην Κριστόλου του τον εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης συνέβαλαν σημαντικά με τα σχόλιά τους. Να αναφερθώ σε ορισμένα εξ αυτών. Και ασφαλώς ε, περιμένω και τις τροπολογίες σας και είμαι ανοιχτό στη συνεργασία μαζί σας με όλους τους κοιόδης και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Σε ό,τι αφορά την κυρία Μερέσ. Συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι αφορά τη σύνταση του EFRS και της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης. Είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά το ρόλο του IFRS 9 κτλ. Σε ό,τι αφορά την πρόταση τώρα, για να μην γίνει η παράταση χρηματοδότηση της ΕΦΡΑΓ, μέχρι ότου υπάρξει μια νέα ε, έκθεση για την πρόοδο της μεταρρύθμισης. Και αυτό γιατί, γιατί έχουμε μια σχετική έκθεση. Και αν καθυστερήσουμε να πούμε στην ΕΦΡΑΚ ότι θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση για το 2016-2020, αυτό θα θέσει την ΕΦΡΑΚ σε μια θέση δύσκολη. Θα αναγκαστεί να πει σε κάποιους υπαλλήλου ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να τους ε, απασχολεί γιατί δεν θα υπάρχει σίγουρη χρηματοδότηση. Θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό, θα το συζητήσουμε και με την Κομισιόν και με την ίδια την Εφράγκα. Τι είδου πληροφορίε τώρα θέλουν να έχουν οι συνάδελφοι επιπροσθέτω ε, προς την έκθεση πρόοδου που υπάρχει σε ό,τι αφορά την, ε, τις εφαρμογές των προτάσεων Μάιστατ της ΕΦΡΑΓ, των συστάσεων Μάιστατ. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι τα σχόλια ήταν πολύ σημαντικά για το θέμα που έθεσε ο συνάδελφος του ΙΣΙΑ ή ο κ. Καμάλ που είναι και Ας Ασφαλώς πρέπει να πω ότι συμφωνώ με πιο πολλά εξ αυτών. Και πάλι έχω μία αμφιβολία σε ό,τι αφορά την εκ νέου μελέτη του IFRS 9 κατά τη διάρκεια της κρίσης. Φυσικά έγιναν πολλές σχετικές μελέτες, ακαδημαϊκές, επαγγελματικέ και το καθεξής. Και ως τώρα φαίνεται ότι το πόρισμα είναι ότι ο αντίκτυπος του IFRS 39 ήταν μεγάλος. Ξέρουμε τι έγινε στον τραπεζικό τομέα, αλλά είναι ασαφές ποιος ήταν ο ρόλος του IFRS 39 κατά τη διάρκεια της κρίσης. Χαίρομαι επίσης και ευγνώμονω την Άλντα για τη συνεργασία. Ευχαριστώ και τους υπόλοιπους συναδέλφους. που έθεσαν το θέμα της σύγκρουσης για να αποφευθεί το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων σε ό,τι αφορά τα θεσμικά όργανα. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Κίγκολτ και τους πράσινους, που είναι μάλιστα ο κύριος Κίγκολτ και πρόεδρος και σχεδόν της ομάδας εργασίας. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα σχόλια για τα θέματα διακυβέρνηση. και ιδιαίτερα ό,τι αφορά το Εποπτικό Συμβούλιο. Συμφωνώ απόλυτα ότι ίσως αυτό το Εποπτικό Συμβούλιο θα πρέπει να διδραματίζει και ρόλο θεματοφύλακα, αλλά να δούμε κατά πόσον αυτό συνάδει με την αρχή της ανεξαρτησίας του ESB αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε με όλους τους συναδέλφους και ίσως θα ξέρετε ότι το Ίδρυμα IFRS βρίσκεται υπό αναθεώρηση κατά πέντε χρόνια. Κάθε πέντε χρόνια, σύμφωνα με τον κανονισμό, προβλέπεται αναθεώρηση του Ιδρύματος. Και εδώ ο Πρόεδρος μου ζητά ευγενικά να ολοκληρώσω. Ασφαλώς θα λάβουμε υπόψη και την έκθεση Τελαροζιέ και θα δούμε τι ακριβώς ε, προβλέπει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συζητήσεις. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε τον εισηγητή, ευχαριστούμε τους κοιόδης, ε, το χρονοδιάγραμμα είναι το εξή. προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών είναι η 1η Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι, εξέταση των τροπολογιών στις 22 Μαρτίου, ψηφοφορία στην εικόνα. 25 ή 26 Απριλίου στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. First vote is uh, on Executive Director, but before that we... Πρώτα θα μιλήσουμε για τον... Uh, καταρχάς θα πρέπει να ελέγξουμε το ηλεκτρονικό μας σύστημα, το σύστημα ψηφοφορίας. Η γραμματεία είναι έτοιμη. Λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για ηλεκτρονικό τσεκ, ηλεκτρονικό έλεγχο. Ο έλεγχος στο τεστ δεν είναι μυστική ψηφοφορία βέβαια. Λοιπόν, ένας ακόμα πρέπει να ψηφίσει. Τέλος της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Θέτουμε σε ψηφοφορία τώρα την πρόταση έγκρισης. Είναι πρόταση του αρμόδιου εισηγητή μετά από την κλεισμένων των θυρών ανταλλαγή απόψεων για το διορισμό του κυρίου Παρέντε ως εκτελεστικού διευθυντή της ΕΑΕΣ για πέντε χρόνια. Ψηφίζεται. Τέλος της ψηφοφορίας 47 υπέρ, 1 κατά, 8 αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν για τον κύριο Παρέντε της Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Περνάμε τώρα στις τρεις εκθέσεις γνωμοδοτήσεις μάλλον, προτάσεις γνωμοδοτήσεων του κυρίου Φέρμπερ για την απαλλαγή των τριών αρχών. Καταρχάς, European Banking Authority, παράγραφος 1, αρχικό κείμενο, ποιοι είναι υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτεί 3 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 4 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 με μια προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 δεν ψηφίζεται γιατί έχει καταπέσει 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο Α, για μια στιγμή λέει ο πρόεδρος. 9 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 13 έχει καταπέσει το αρχικό κείμενο. Α, δεν είναι απαραίτητο. Τότε η 17 έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε τη 18. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 19. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίφτεται. 20. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 22. Υπέρ, κατά, αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά 23 η 21 έχει καταπέσει δεκτή 23 λέει ο πρόεδρος 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 29 τέλος της ψηφοφορίας δεκτή 29 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή το σύνολο τροπολογημένο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζεται ηλεκτρονικά. «43 υπέρ, 3 κατά 9 αποχές δεκτή η πρόταση. Συγχαρητήρια στον εισηγητή». Τώρα θα μιλήσουμε για την ΑΙΟΠΑ. Παράγραφος 1 του αρχικού υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές δεκτό 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Παράγραφος 4 αρχικό υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17. Πηγαίνουμε στη 17. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 18. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 21. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 22. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές Δεκτή η ίδια πλειοψηφία. Τροπολογημένο κείμενο τώρα ψηφίζεται ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. 44 υπέρ, 3 κατά 10 αποχές. Και περνάμε τώρα στην ΕΣΜΑ. Αρχικό κείμενο Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 5 με προφορική υπέρ κατά αποχές δεκτές, 6, 7 μάλλον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 8 εν, υπέρ κατά αποχές δεκτή, 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο στην 4, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 10, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 11, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 17, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 14, υπέρ, 18, όχι 14, 18, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 21 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 30 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 25 υπέρ, Α, όχι, το 27. Ψηφίζουμε το 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή 27. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή το απολογημένο το κείμενο ηλεκτρονική ψήφος Τέλος. Συγχαρητήρια στον εισηγητή για τη σκληρή δουλειά που έκανε. Και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ασφάλισης Καταθέσεων απλοποιημένη διαδικασία εδώ έτσι, για την, το Ευρωπαϊκό Σύστημα ε, Ασφάλισης Καταθέσεων. Okay, so uh, it is the first exchange of view on the. Πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Όπως ξέρετε, η πρόταση της Κομισιόν είναι αυτή για την ασφάλιση των καταθέσεων και δίνουμε το λόγο στον κύριο ε, στην κυρία Ντελάνγκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Σήμερα λοιπόν έγινε μια, γίνεται μια απόψεων για ένα θέμα το οποίο μας έχει ε, πολύ. Κάποιοι συνάδελφοι ήθελαν να έχει ήδη γίνει η πρόταση, αν ήταν δυνατόν χθες και άλλοι συνάδελφοι δεν θα θέλουν να έχει γίνει ποτέ η πρόταση αυτή. Φυσικά υπάρχουν διαφορές και μεταξύ των ομάδων, αλλά φαντάζομαι ότι θα ακούσουμε τις διαφορετικές απόψεις σήμερα το απόγευμα σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Εγώ ήλθα λοιπόν ως ηγήτρια σε πρώτη φάση για να ακούσω. Νομίζω ότι αυτό που μας απασχολεί, πολλούς από εμάς, είναι το τι γίνεται στην Τραπεζική Ένωση και η, το οικοδόμημα με τρεις πυλώνες. Ε, εποπτεία, ε, ασφάλιση των ε, καταθέσεων, ότι αυτό μας εξυπηρετεί. Οι πιο θεωρούμε ότι ακριβώς αυτοί οι τρεις πυλώνες θα υπήρχαν σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια όμως να σκεφτούμε μόνο σε ακαδημαϊκούς όρους για την πρόταση αυτή και η πρόταση αυτή έρχεται μια χρονική στιγμή και σε ένα πλαίσιο όπου ε, χαρακτηρίζεται από έλλειψη εμπιστοσύνης και στις αγοράς και μεταξύ των χωρών. Δεν είναι τόσο ήσυχα τα πράγματα όσο θα θέλαμε και στην παρούσα φάση ενδεχομένω να υπάρχουν και ερωτηματικά σε ό,τι αφορά το σεβασμό του υφιστάμενου πλαισίου της Τραπεζικής Ένωσης. Τι γίνεται με τον Μπέιλιν, για παράδειγμα. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε στη θεωρία αυτό Τώρα στην έννοια αυτή υπήρχε και το σημαντικό θέμα του moral hazard, του ηθικού κινδύνου την προηγούμενη περίοδο και αναρωτιωστόμαστε κατά πόσον ε, υπάρχει επαρκή σεβασμός του πλαισίου προκειμένου να το επεκτείνουμε. Να ξεκινήσω όμως ε, από την αρχή και να θέσω το ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί μια επιτροπή η οποία δεν κάνει ποτέ προτάσεις χωρίς μελέτη αντικτύπου σε ένα τόσο σημαντικό θέμα και τόσο αμφελιγόμενο έρχεται και δεν κάνει μελέτη αντικτύπου. Καταλαβαίνω ότι υπήρχε πάρα πολλά να κάνει το 2010. Υπήρχε και μία άλλη πρόταση και τότε δεν ε, υπήρχαν πολλά τέτοια δεδομένα και θα έπρεπε, μάλλον ε, αναγκαστικά δουλέψαμε με εικαζόμενα πόσα. Τώρα όμως έχουμε τέτοια αριθμητικά στοιχεία. Γιατί δεν κάναμε μία μελέτη αντικτύπου λοιπόν πια. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο ήθελα να το θέσω και το οποίο είναι σημείο κλειδί στο φάκελο αυτό η σύνδεση μεταξύ μείωσης και κατανομής του κινδύνου. Σε πολλά θέματα το έχουμε θίξει το θέμα αυτό, κατά πόσον ε, θα μπορεί το ένα να αντικαταστήσει το άλλο, κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχουν και τα δύο και υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για το θέμα αυτό και ξέρω ότι κάποιοι ισχυρίζονται ότι φτάνει πια η κατανομή του κινδύνου και ότι φτάνει και η μείωση του κινδύνου και αρκετά έχουμε κάνει για να μοιάσουμε τον κίνδυνο, αλλά στην πράξη, και εγώ την πράξη θέλω να κοιτάω, όχι μόνο τι γίνεται στα χαρτιά, στην πράξη τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Η κυρία Κιούνιχ από τον ΕΣΜΠ μας είπε ότι ο ορισμός των σχετικών όρων θα γίνει στα τέλη του έτους και ούτω καθεξής. Άρα η σχέση μεταξύ των νομοθετικών κειμένων και μια ανακοίνωση για την μείωση του κινδύνου θα είναι βασικό ζήτημα στο φάκελο αυτό και θα πρέπει τα... κατά πόσον αυτά τα δύο θα πρέπει να εναρμονιστούν το μεν με το δε και να ελέγχονται και τα δύο για να δούμε κατά πόσο ε, είναι απαραίτητα αυτά για την κίνηση αλλά και για τις μετέπειτα φάσεις του φακέλου αυτού. Και γι' αυτό λοιπόν κύριε Πρόεδρε Θέλω να υπάρξει ένα σαφή σύνδεσμο και νομίζω ότι δικαίω μεταξύ τη νομοθετική πρόταση και τη συζήτηση για τη μείωση του κινδύνου. Σα ε, προειδοποιώ ότι δεν θα πρέπει να συνδεθεί ο φάκελο με άλλα θέματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν τίποτα με αυτό. Και σας προειδοποιώ ότι θα χρειαστούμε χρόνο για να καταλήξουμε στα συμπεράσματα. Αν σκοπός μας είναι να μην συνδέσουμε άσχετα θέματα προκειμένου να βιαστούμε θα πρέπει να σας πω ότι εγώ ε, η συγκεντρία δεν ε, με πείθετε. Δεν πρέπει να βιαστούμε, πρέπει να είμαστε ενδελεχείς και να εξετάσουμε το περιεχόμενο προκειμένου τελικά να μπορέσουμε να κάνουμε τα σωστά βήματα με ευρεία συνένεση. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα, δεν είναι ένα θέμα το οποίο θέλουμε να περάσει οριακά στο Κοινοβούλιο. Αυτά είναι τα εισαγωγικά μου σχόλια. Επαναλαμβάνω ότι ήρθα εδώ για να ακούσω βασικά. Έδωσα κάποια ενάρσματα για τη συζήτηση και είμαι σίγουρη ότι θα ακούσω πολλά και διαφορετικά σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Η κυρία Φερέιρα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια, την κυρία ε, Στελαντελάγκη, για αυτή την πρώτη της ε, εισήγηση. Πιστεύω πως πρόκειται για μια υπόθεση όπου οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα ζητήματα ε, δηλαδή να πούμε γιατί χρειαζόμαστε αυτό το σύστημα, πότε και έπειτα το περιεχόμενο. Θέλουμε ε, σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση να το κάνουμε ή καλύτερα θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή στα πρώτα δύο γιατί λέμε ότι το περιεχόμενο θα εξεταστεί στις επόμενες συνεδριάσεις. Τώρα, γιατί χρειαζόμαστε ένα τέτοιο σύστημα. Εγώ πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να θυμίσουμε ότι εφόσον υπάρχει η Τραπεζική Ένωση που συμφωνήθηκε από την Ένωση βασικό της στόχο είχε να σταθεροποιηθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας και να κοπεί ο δεσμός ανάμεσα στις τράπεζες και τις, τα κράτη. Και τα είχαμε συμφωνήσει με σε ένα κοινό βιβλίο, CRD, BRD, ένα σωρό νομοθετήματα τα οποία εμείς εκπονήσαμε όπου οι τρεις πυλώνες ήταν κοινή εξυγίαση και νέα συστήματα εγγυήσεων των καταθέσεων. Θεωρήσαμε πως αυτός ο πυλώνας θα έπρεπε να εξεταστεί από κοινού από τη στιγμή που θα είχαμε τους κοινούς κανόνες για την αθεώρηση. Η Τραπεζική Ένωση λοιπόν εξασφαλίζει την κοινή εφαρμογή ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των κανόνων και κατέστησα σαφές εξ αρχή ότι μπαίναμε σε χαρτογράφητα νερά και ότι θα χρειαζόταν εδώ μελέτη επιπτώσεων περισσότερο ακόμη από ότι με το bail-in και την εξυγίανση και για άλλα στοιχεία που υποτίθεται ότι σταθεροποιούν όλη, όλο αυτό το σχέδιο. Η Τραπεζική Ένωση ακολουθεί αυτή την κοινή εφαρμογή. Θα πρέπει τώρα να θυμόμαστε ότι από τον Νοέμβριο του 2014 η ΕΚΤ μέσω του νέου μηχανισμού είναι η εποπτική αρχή και έχουμε και τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης με το ενιαίο ταμείο εξυγίανσης και όλα αυτά ξεκίνησαν ήδη από την πρώτη πρώτου του τρέχοντος. Στην πράξη έχουμε χωρίσει τις δύο φάσεις. Δύο φάσεις που είναι ο μηχανισμός εξυγένσης και το σύστημα ασφάλισης καταθέσεων. Πιστεύω πως είναι σημαντικό να θυμίσουμε εδώ ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε σε σχέση με την ασφάλιση των καταθέσεων, δηλαδή το τρίτο πυλώνα, ήδη έπρεπε να έχει γίνει και το υποσχέθηκε το Συμβούλιο και η Κομισιόν και συγκεκριμένα θυμάμαι ότι ο προηγούμενος πρόεδρος ο Ντουράου Μπαρόζο δήλωσε δημόσια και μάλιστα στους Financial Times ότι αναμφίβολα έπρεπε η Τραπεζική Ένωση να συμπεριλαμβάνει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων. Και στην έκθεση των πέντε προέδρων αναφέρθη ως ο τρίτος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης. Ε, the banking union so uh, is uh, is consisting of three pillars, and I don't think we should uh, discuss this any longer. Um, and we should just move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 Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις διαφορές ε, είχαμε ότι στο ETFC η αγγίση των, ασφαλί... καταθέσεων ήταν ε, το πρώτο βήμα για την εξασφάλιση τραπεζικής ένωσης και μετά υπήρχε η... Ε, ο άλλος πυλώνας. Εμείς λοιπόν εδώ πρέπει γρήγορα να ενεργήσουμε ε, πρέπει να υπάρχει ε, ένα γεφύρωμα των χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων που πρέπει να στηρίξουν ε, το ενιαίο Ταμείο Εξυγίνησης και να μπορέσουμε έτσι να φτάσουμε σε πλήρη ανακεφαλοποίηση. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια κοινή πιστωτική γραμμή και εθνικές πιστοτικές γραμμές ώστε να λειτουργεί το Ταμείο. Η πιστοτική γραμμή από τον ESM που υποσχεθήκαμε από το 2010 λείπει, εξακολουθεί να λείπει και βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν όσο γίνεται πιο σύντομα. Πότε, ήδη το απάντησε αυτό, πιστεύω απλώς και κάνω έκκληση στους συναδέλφους ότι επειδή αυτό το κοινοβούλιο ήταν τόσο δραστήριο και ενεργό στην κατασκευή της Τραπεζικής Ένωσης, δεν θα πρέπει να δώσει το μήνυμα ότι μπορούμε εδώ να χαλαρώσουμε και να χασομερίσουμε το Συμβούλιο ή εξετάζει πολύ σοβαρά το περιεχόμενο της πρότασης της Κομισιόν και την ουσία του προβλήματος. ορίζω την πρόταση που ήρθε από την Κομισιόν, αν και δεν είναι η αρχική της πρόταση. Είναι ωστόσο μια πολύ ενδιαφέρουσα βάση για να εργαστούμε από αυτή και θα πρέπει να σκεφτούμε το χρονοδιάγραμμα και μάλιστα να επιταχύνουμε σε σχέση με αυτό το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται. Δεν είναι αρκετά γρήγορο δεν μας κάνει και τη το τελικό όραμα, τι θέλουμε να πετύχουμε. Και από αυτού αναμφίβορα χρειάζεται ένα στοιχείο σταθεροποίησης από αυτά που λείπουν. Χρειάζεται ένα στοιχείο σταθεροποίηση από τα δύο που λείπουν. Και να είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε για τις λεπτομέρειες, αλλά και πάλι όσο γίνεται πιο σύντομα και χωρίς να αφήσουμε το Συμβούλιο να ηγηθεί. Γιατί ήμασταν ανέκαθαν εξαιρετικά δραστήριοι και κατά κάποιο τρόπο προς εμάς στρέφονται οι πολίτες για την ε, σε αυτό το περίπλοκο κόσμο για 130.000 καταθέσεις και γι' αυτό μιλάμε το πράγμα. Αυτά τα στοιχεία είναι λοιπόν απαραίτητα για να ενισχύσουμε και να παρέχουμε ένα μήνυμα εγγύησεων στην ε, χρηματοπιστωτική αγορά. Να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Κάνατε μια εξαιρετική εισαγωγή. Θέλω να σας ευχαριστήσω και ε, για την ε, πρόταση χρονοδιαγράμματος. Βρίσκουμε ότι είναι εξαιρετική. Εμείς θέλουμε να είμαστε επικοδομητικοί πάνω σε αυτό το θέμα σαν ομάδα του ECR. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για όλους. Θα απαιτηθεί πολύ σκληρή δουλειά για τη σημερινή συζήτηση θα αναφερθώ σε ορισμένες γενικές γραμμές. Για την πολιτική μας ομάδα κάθε πρωτοβουλία που έχει σαν στόχο να προστατεύει τους καταθέτες, να προωθεί την χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο να εξετάσουμε. Στην τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση είδαμε πως πήγαν τα πράγματα, δεν έχουμε ακόμα συνέλθει είναι υπερχρεωμένα τα πιστοτικά ιδρύματα και τα κράτη-μέλη και αυτό εμποδίζει την, την οικονομική ανάπτυξη. Κατανοώ την λογική σας για το σύστημα εγγυήσεων, το σύστημα ασφάλισης μάλλον. Είναι ένα σύστημα το οποίο όμως είναι ευάλωτο σε μεγάλα συστημικά σοκ. Οποιοδήποτε πάντως ευρωπαϊκό πρόγραμμα ασφάλισης θα πρέπει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συστημική σταθερότητα του συστήματος ε, στο σύνολο της Ευρώπης αλλά και σε επιμέρους σταθεροποίηση των εθνικών συστημάτων και όχι να μεταφέρει το κόστος και τον κίνδυνο από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Αυτό θα ήταν ανεύθυνο και δεν θα υποστηριχθεί από την εκλογική μου περιφέρεια. νομίζω ότι δεν υπάρχει μία παράγραφο στην πρότασή σας που να μην δημιουργεί συζητήσεις. Αυτό ε, είναι καλό γιατί θέλουμε εμείς να δημιουργήσουμε κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οπότε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την παρούσα κατάσταση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν με έχει πείσει ότι όλα πηγαίνουν καλά στον τομέα αυτό. Κοιτάξτε τι συμβαίνει στην Ιταλία. Απαιτείται η συζήτηση να γίνει και με διαφορετικό τρόπο για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο και όχι να περάσουμε απευθείας στην φάση της κατανομής του κινδύνου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο ζητάμε τώρα είναι να σώσουν οι βόρειες τράπεζες, οι τράπεζα στις βόρειες χώρες, ε, τους, τις Έλληνες καταθέτες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται μεγαλύτερη συζήτηση. Για να προστατευτούν οι ευρωπαϊκές καταθέσεις πρέπει να αυξηθεί η συστημική σταθερότητα και να μειωθούν οι κίνδυνοι μιας μεγάλης πιστοτικής κρίσης στο μέλλον. Δεν θα πρέπει να τα όλα με όλα τα άλλα επίπεδα, αλλά υπάρχουν μεμονωμένα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πολλά έχουν ήδη γίνει για την αύξηση και τη βελτίωση της σταθερότητας. Πολλοί πιστεύουν βέβαια ότι υπάρχουν υπερβολικοί διακανονισμοί και ρυθμίσεις και ότι είναι το σύστημα ιδιαίτερος γραφειοκρατικό. Υπάρχουν και τα μη συμβατικά μέτρα από τους κεντρικούς τραπεζίτες. Ο κύριος Ντράγκη μας επισκέφθηκε επανειλημμένα και αυτά τα μη τυπικά, μη παραδοσιακά μέτρα αυξάνουν τον κίνδυνο της ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Αυτό δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Και όπως είπε και η συγγήτρια, συμφωνούμε μαζί της για το ότι η επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να μην γίνει μια νέα μελέτη επιπτώσεων ή να μην υπάρξει μια επικαιροποίηση της προηγούμενης. Αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε ζητηθεί και στα πλαίσια της εκθέσεως των πέντε προέδρων. Συμφωνώ λοιπόν με πολλούς από τους συναδέλφους σε αυτή την αίθουσα που πιστεύουν ότι αυτά τα οποία περιλαμβάνονται ε, στην ε, έκθεση των πέντε προέδρων δεν πρέπει να εξαιρούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το να κάνει την σωστή δουλειά την οποία καλείται να κάνει. Το θέμα της εκτίμησης των επιπτώσεων και την αξιολόγησή τους είναι κάτι το βασικό που θα έπρεπε να κάνει η Επιτροπή. Όταν βλέπω την έκθεση του 2010, το σημείο 7 και μετά το σημείο 11, λέγεται ότι η διασυνοριακή συνεργασία της ε, ε, Γενικής Διεύθυνσης της Αρμόδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις αρμόδιες εθνικές αρχές καλύπτει τέσσερις σελίδες. Τέσσερις σελίδες σε μια έκθεση 150 ε, σελίδων συνολικά. Λίγα έχουν γίνει και πολλά μένει να γίνουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα κλείσω εδώ ίσως με κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με τις ανάγκες οι οποίες θα πρέπει να οριστεί ότι υπάρχουν. Πρώτον, ε, μελέτη επιπτώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει ε, σε τέτοιες μελέτες ήδη από τον Απρίλιο. Να δούμε επίσης τι, ε, πώς θα επηρεάσει την πραγματική οικονομία και τον πιστοτικό φυσικά τομέα. Τα λεγόμενα legacy cost, δηλαδή ό,τι έχει απομείνει σαν κόστος για τις μικρές τράπεζες από την προηγούμενη κρίση και πώς επίσης θα μειωθούν και οι περιπτώσεις δεοντολογικού κινδύνου τα λεγόμενα moral hazard cases. Λοιπόν, ε, κλείνοντας ευχαριστώ την εισηγήτρια, είναι σωστή η αντιμετώπιση σας, ευχαριστώ επίσης και για την σωστή πρόταση χρονοδιαγράμματος που θα σε μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε το θέμα με σοβαρό τρόπο και να του δώσουμε και την προσοχή που σίγουρα του αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Η σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτριά μας, ε, όντως, που ήδη μας ε, ε, κάλεσε εδώ για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Εγώ συμφωνώ με κάποια από αυτά που ήδη υπόθηκαν. Τρίτη ο πυλώνα τη Τραπεζική Ένωση. Αυτό υπενθυμίστηκε στην έκθεση των πέντε Προέδρων. Θα πρέπει να διαμαρτυρόμαστε. Ξέρουμε ότι ορισμένε αποφάσει του Συμβουλίου μένουν νεκρό γράμμα. Εδώ όμω η συλλογική μα αξιοπιστία διακυβεύεται και βεβαίω θα πρέπει να ε, επιμείνουμε στο δικαίωμα πρωτοβουλίας Κομισιόν. Ε, στην οδηγία που υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2014 σημειώνουμε ότι λέει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να υποβάλει νέα πρόταση το αργότερο τον Ιούλιο του 2019. Οπότε τύπης είμαστε εντός των χρονικών ορίων. Στην επιτυχία είναι ένα θέμα περίπλοκο δεν θα πρέπει να το αποκρύψουμε, ε, όχι μόνο πολιτικό ευαίσθητο, αλλά και κυρίως αυτό που θα πρέπει να μας καθοδηγήσει εδώ. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ακριβώς τι χρειαζόμαστε δεδομένων των μέτρων που εμείς ήδη λάβαμε. Μετά από τη δημιουργία ενός συστήματος εποπτείας και εξηγήσεις, η καθάριση πρόκειται για ένα συμπλήρωμα που έρχεται φυσιολογικά γιατί εδώ είμαστε συνδεδεμένοι με την ύπαρξη μιας εσωτερικής αγοράς με, αν είναι δυνατόν, κατανομή κεφαλαίων που να ξεπερνά τα σύνορα, να είναι διασυνοριακή. Τώρα, για την ένταση, το ρυθμό μπορούμε να το συζητήσουμε. Είναι προφανές ότι δεν υπήρξε μελέτη αντικτύπου. Ε, πρέπει όμως να προσέξουμε τι σημαίνει αυτό για ε, τον τραπεζικό τομέα και για τη διαφοροποίηση του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη ώστε να μην είναι αυτό εις βάρος του τραπεζικού τομέα, αλλά ταυτόχρονα να δοθεί εγγύηση για όλους τους αποταμιευτές, όλους γιατί πιστεύω ότι και εδώ υπάρχει μια διαφορά βορρά-νότου που είναι λυπηρή. Εδώ ε, νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για όλους και να είναι όλοι σωστά και κατάλληλα προστατευμένοι. Το σύστημα τώρα ασφάλισης ε, πλήρους ασφάλισης ε, και πώς ε, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα, να σημειώσω ότι ακόμα δεν έχουμε γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι πολύ σημαντική εδώ. Η Εστέρ καλά έκανε και προέβλεψε και ακροάσεις. Χρειάζεται να το συζητήσουμε με διάφορα φορείς και να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι συνθήκες της ε, συγκέντρωσης των κονδυλίων, όχι μόνο ρυθμός, αλλά και πώς θα προχωρήσουμε. Τώρα, για τα άλλα τα ζητήματα Όλα είναι μεταξύ τους συνδεδεμένα, αλλά συμφωνώ με την ιδέα ότι θα πρέπει ίσως να μείνουμε σε ένα σχετικά περιορισμένο πεδίο. Βέβαια, ανάλογα με το θα πρέπει να δούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο να αξιολογούμε το, τα, το χρέη, τα χρέη τα κρατικά ε, θα πρέπει να δούμε επίσης ε, τους κανόνες πτώχευσης ε, σε σχέση με την Τραπεζική Ένωση και επίση είναι σημαντικό να βελτιωθεί η διακυβέρνηση των τραπεζών. Δηλαδή να υπάρχουν προληπτικά και ποιοτικά μέτρα που μπορεί να μειώσουν του κινδύνου πέρα από την απλή μείωση τη συσχέτιση ανάμεσα στο κρατικό τομέα και στι τράπεζε. Είχα υποβάλει σχετικέ τροπολογίε εξάλλου και παλιότερα. Τελευταία μου παρατήρηση που σχετίζεται με την πρόταση πρωτοβουλία που πρόσφατα κάναμε είναι σημαντικό να δούμε τι κάνει η Επιτροπή της Βασιλείας για αυτό το θέμα, ώστε η δική μας νομοθεσία να ενταχθεί σε μια γενική προσέγγιση, αν και φυσικά είμαστε ανεξάρτητοι στις δικές μας αναλύσεις. Χαίρομαι λοιπόν που θα συνεργαστώ με μια ομάδα εισηγητών εξαιρετικά ψηλή ποιότητα και φυσικά το δικό μου γραφείο θα είναι πάντοτε ανοιχτό για να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε. Δεν είμαι απόλυτη τώρα για το χρονοδιάγραμμα, δεν θα ήθελα να καθυστερήσουμε, αλλά από την άλλη πλευρά να έχουμε και τον κατάλληλο χρόνο, ειδικά στι χώρε όπου γίνεται έντονη δημόσια συζήτηση, να καθησυχαστεί ο κόσμο, να δούμε όλα τα θέματα, να έρθουμε σε επαφή με όλους τους φορείς, γιατί το θέμα δεν είναι ε, να επιβάλλουμε κάτι, είναι να πείσουμε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Δημήτρης Παπαδημούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις εισαγωγικές της παρατηρήσεις. Άκουσα με ενδιαφέρον και τους κοιόδης εισηγητές που προηγήθηκαν. Θα προσπαθήσω όσο πιο απλά γίνεται να σας περιγράψω τη σκοπιά από την οποία βλέπω εγώ τα πράγματα και η πολιτική μου ομάδα το θέμα που συζητούμε, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύης Καταθέσεων, έχει πολλές δυσκολίες και πολλές τεχνικές πλευρές και χρειάζεται να το συζητήσουμε. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και ένας από τους τρεις πυλώνες μιας συμφωνημένης, αποφασισμένης, σχεδιασμένης τραπεζικής ενοποίησης που σημαίνει ότι εάν δεν προχωρήσει ο τρίτος πυλώνας και έχουμε μία παραπομπή του στις καλένδες, τότε θα προσθεθούν κίνδυνοι, θα αυξηθεί η αστάθεια και από αυτό θα ζημιωθούν όλοι. Όχι μόνο το τραπεζικό σύστημα, αλλά όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Γι' αυτό είμαι κατηγορηματικά αντίθετος στην προσέγγιση αυτού του δύσκολου θέματος με διαιρετική προσέγγιση. βοράς εναντίον νότου. Λάθος προσέγγιση. Όπως επίσης δεν μπορώ να συμφωνήσω με μια φράση, αν την άκουσα καλά από τη διερμηνία, ενός σκιώδους συγητή που λέει ότι όλη αυτή η πρόταση της Κομισιόν είναι για να προστατευτούν οι ελληνικές τράπεζες νομίζω ότι πολύ απέχει η Κομισιόν από το να κατηγορείται για κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μέτρα που να ενισχύουν τη σταθεροποίηση και την πρόοδο στο τραπεζικό σύστημα που να βοηθήσει την ανάπτυξη και την ανάκαμψη. Και ήδη αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, η Κομισιόν έκανε τρία χρόνια για να παρουσιάσει την πρότασή της. Και η πρόταση της Κομισιόν που κατά τη γνώμη μου είναι μια καλή βάση για συζήτηση, μακριά από το να είναι τέλεια, προβλέπει και μια μακρά διαδικασία εφαρμογής με στάδια που καταλήγουν μέχρι το 2024 για την ολοκλήρωσή της. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι αν στο θέμα αυτό προχωρήσουν μόνο οι δύο από τους τρεις πυλώνες θα έχουμε μια αναπηρία και μια αναποτελεσματικότητα στην τραπεζική ενοποίηση. Επειδή δεν θέλω να μακρηγορήσω, θα θέλω να σας πω σε αυτή την πρώτη συζήτηση που έχει αναγκαστικά γενικό και αναγνωριστικό χαρακτήρα, ότι κατά τη γνώμη μου το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να παίξει έναν ενεργό επικοδομητικό ρόλο στην διαμόρφωση αυτού του τρίτου πυλώνα και να μην περιμένει απλώς να δει προς τα που θα φυσήξει ο καπνός στη συνεδριάση του Συμβουλίου ή αν θα βγει καπνός. Δεν ταιριάζει στο Ευρωκοινοβούλιο ο ρόλος ενός ευρωπαϊκού θεσμού που απλώς περιμένει να δει προς τα που θα πάνε τα πράγματα στο Συμβούλιο για να δούμε και εμείς τι θα πούμε μετά. Χρειαζόμαστε χρόνο και το υποστήριξα και στην συνάντηση των σκιωδών εισηγητών για να κάνουμε όλες αυτές τις δημόσιες ακροάσεις, να εξετάσουμε το θέμα από όλες τις πλευρές, χρησιμοποιώντας και τη γνώμη των ειδικών. Είμαι κατηγορηματικά υπέρ μιας ουσιαστικής συζήτησης, αλλά είμαι κατηγορηματικά επίσης εναντίον της παραπομπής του θέματος στις ελληνικές καλένδες, στις αρχαίες, στο όνομα των υπαρκτών δυσκολιών. Δεν μπορούμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να έχουμε μία προσέγγιση για τα θέματα της ενοποίησης αλλά κάρτ. Να τρέχει η ενοποίηση σαν λαγός όταν πρόκειται να υπηρετηθούν συγκεκριμένες προτεραιότητες και σκοπιμότητες και σε άλλα θέματα να πηγαίνουμε με βήμα σημειωτών ή και προς τα πίσω. Είναι δική μας ευθύνη εδώ να συζητήσουμε και να συνθέσουμε απόψεις γιατί συμφωνώ με την ε, εισηγήτρια ότι όσο πιο ευρία είναι η συνένεση στην οποία θα καταλήξουμε ως Ευρωκοινοβούλιο τόσο αποτελεσματικότερη δουλειά θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λάμπερτ. Πρόεδρε. Και πάντα χαρά μου να σας βλέπουμε. Έστερ, πρώτη φορά θα συνεργαστούμε μαζί. Προσβλέπω σε αυτή τη συνεργασία. Ήξερα από τον προχάτοχό σας, ήταν καλή η συνεργασία. Ελπίζω να τα πάμε εξίσου καλά. Είπατε κάτι στα εισαγωγικά σα σχόλια ότι το θέμα αυτό είναι πολύ αμφιλεγόμενο και προκαλεί μεγάλο διχασμό και μεταξύ πολιτικών ομάδων αλλά και στο εσωτερικό πολιτικών ομάδων. Εγώ δεν ξέρω αν καφιέμαι, αλλά στο θέμα αυτό πρέπει να σας πω ότι η πολιτική μας ε, ομάδα είναι ενωμένη και μιλώ για τους, και για τους Γερμανούς πράσινους. Στα γερμανικά κυρίως, ε, Λάμπερτ. Παρά το γεγονός ότι δεν είμαι Γερμανός, μας ενώνει η ιδέα ότι ναι, χρειαζόμαστε αυτόν τον τρίτο πυλώνα της ε, Τραπεζικής Ένωσης και συμφωνώ με την άποψη όσων διατείνονται ότι ο πυλώνας αυτός έχει μείνει πίσω πολύ καιρό και εγώ θα ήθελα να έχει δημορφωθεί πιο νωρί, αλλά εδώ βρισκόμαστε εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει νόημα να κλαίμε για τα σπασμένα, να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε. Βάσει τη πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πιστεύω, όπω είπε και ο Δημήτριο, ότι κινείται προ τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι τέλεια, εντάξει και Σάντερ ενδεχομένω να μην υπήρχε πλήρη μελέτη αντικτύπου, αλλά όποτε γίνεται πλήρη ε, μελέτη αντικτύπου θα πρέπει να δούμε και να γίνεται και μελέτη αντικτύπου τη μη δράση. Τι θα γίνει άμα καθυστερούμε, άμα αργούμε. Και ναι, μπορούμε να χτενίσουμε την ανάλυση και να κοιτάξουμε τις λεπτομέρειες, αλλά αυτό να μην είναι επίφαση για την αδράνειά μας, γιατί υπάρχει και κόστος της αδράνειας και σύμφωνο μαζί σας Έστερ ότι δεν θα πρέπει να τα μπλέκουμε όλα, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η ιδέα σε ό,τι αφορά της μείωση και της προστασίας κινδύνου. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και στις δύο πλευρές. Δεν λέω ότι θα πρέπει να γίνει σύνδεση με πράγματα που συμβαίνουν εκτός του νομοθετικού κειμένου, Πιστεύω όμως ότι στο εσωτερικό του νομοθετικού κειμένου θα μπορούσαμε να, να μιλήσουμε και για την ε, μείωση του κινδύνου και για την αμοιβοποίηση του κινδύνου. αμοιβοποίηση του κινδύνου. Και πιστεύω για παράδειγμα ότι στον, με τον τρόπο που δομείται τις σύμβολες στο Ταμείο Συμβολών μπορεί να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να δοθούν κίνητρα για τη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών. Ένα παράδειγμα μόνο. Αν πει κανείς ότι το χαρτοφυλάκιο, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το εθνικό χρέος, δεν θα επιτεθούν σε μία χώρα, αλλά θα μετρηθούν, θα κατανεμηθούν σε πολλές χώρες, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα από ότι αν υπάρχει έντονη επικέντρωση σε μια χώρα. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό ενδεχομένω μπορούμε να ε, δώσουμε ένα έναυσμα για τη μείωση του κινδύνου. Και να σας πω ότι ο κίνδυνος είναι παντού. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή για να πούμε το εξής. Αν θέλουμε να υπάρξει αμοιβαιοποίηση των ασφαλίσεων των καταθέσεων, ίσως θα πρέπει να κάνουμε άλλο ένα βήμα για τη μείωση του κινδύνου με αυτό το κείμενο, όχι με άλλα μέσα και μέσα στο κείμενο αυτό θεωρώ ότι έχουμε πολλές ευκαιρίες. Ένα άλλο σημείο που ήθελα να αναφέρω. Όντω, ε, όλη η νομοθεσία εω τώρα ήταν one size fits all, ε, μία λύση για όλου. Ε, με μία τράπεζα κατά νου. Και υποστηρίζω όσου λένε ότι υπάρχουν συστήματα που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά. Δεν θέλουμε τα συστήματα αυτά να σβηστούν με μία μόνο κοντιλιά από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων. Θα πρέπει να προβλέπεται αυτή η διαφοροποίηση με ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέπει κάπως μεγαλύτερη ε, διαφοροποίηση στην εφαρμογή. Θα πρέπει να δούμε και το θέμα του του backstop, γιατί ξέρουμε ότι θα πάρει χρόνο να παραλυθούν οι καταθέσει στα φυσιολογικά επίπεδα. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι εγγυήσει καταθέσεων να είναι αξιόπιστε σε κάθε φάση. Να προσθέσω τώρα κάποιες ε, παρατηρήσει. Ναι, το χρηματοπιστωτικό σύστημα εμπεριέχει πολλούς κινδύνους ακόμα. Παντού. Αλλά στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω κάτι ίσως που να ακουστεί πολιτικό. Αλλά ειλικρινά, ένας από τους βασικούς λόγους που υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι επειδή ποτέ δεν ε, βγάλαμε τα κακά στοιχεία. Ποτέ δεν το ξεκαθαρίσαμε. Στις είπα ενδεχομένω να έχουν ε, πάει και παραπέρα σε ό,τι αφορά την απομάκρυνση των ε, βασικών στοιχείων που είναι αρνητικά. Αλλά υπάρχει ένα ταμπού για τον καπιταλισμό. Ότι ο κόσμο ε, παίρνει λάθο επιχειρηματικέ αποφάσει και υπόκειται τι ζημίε. Υπάρχει αυτή η λάθο αντίληψη. Και αυτό είναι ένα από του βασικού λόγου που καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Δεν θέλαμε να υποστούν τις συνέπειε οι Ιρλανδικές τράπεζε και τελικά τι υπέστησαν οι Ιρλανδοί πολιτέ Το ίδιο με την Ελλάδα και με τον ε, Έλληνα φορολογούμενο και με τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό ήταν ε, σοφό ως κίνηση. Τέλος για το, το χρονοδιάγραμμα. Αν είχα την αίσθηση ότι μια συμφωνία η οποία πραγματικά ιδρύει αυτόν τον τρίτο πυλώνα με αξιόπιστο τρόπο, με ευρεία πλειοψηφία θα μπορούσε να επιτευχθεί γρήγορα, θα την υποστηρίζα. Πραγματικά θα την υποστηρίζα. Ε, σοβαρά το λέω. Αλλά ξέρουμε ότι είναι δύσκολο και αν είχα την αίσθηση ότι ο χρόνος είναι κατά μας, γιατί τώρα ε, σχεδόν έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με μια μικρή προσπάθεια, θα την πετυχαίναμε, θα έλεγα ας κάνουμε αυτή την επιπλέον προσπάθεια. Αλλά θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε μια μπλοκαρισμένη πολιτική κατάσταση. Για να λύσουμε όλους τους ε, κόμπους θα χρειαστεί ίσως χρόνος. Είμαι υπέρ της ταχύτητας, αλλά είμαι και ρεαλιστής παράλληλα. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούμε γρήγορα να πετύχουμε τη λύση η οποία θα, την οποία θα υποστηρίξει μεγάλη πλειοψηφία εδώ πέρα. Και αυτό το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε. Αυτά λοιπόν για τη μελλοντική μας συνεργασία στην οποία και προσβλέπω. Μάρκο ehm. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την γιατί η πρώτη συνάντηση ήταν ενδιαφέρουσα για να μπορέσουμε να θέσουμε τις βάσεις για αυτή τη σημαντική συζήτηση. Δεν το επαναλαμβάνω και εγώ γιατί το είπαν σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι που προηγήθηκαν ότι αν θέλουμε να έχουμε σταθερότητα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε αυτή η διάταξη να υπάρχει γιατί είναι βασικό σημείο ώστε το ε, σύστημα το τραπεζικό να είναι πιο αξιόπιστο ενώπιον των πολιτών και πιο ε, συμπαγές ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει την πραγματική οικονομία. Οπότε οπωσδήποτε αυτή η διάταξη είναι απαραίτητη και μάλιστα έχει και αργοπορήσει. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα δουλεύοντας πάνω σε ένα κοινό σχέδιο εγγυήσεων για τις ε, ε, καταθέσεις να διορθώσουμε και κάποιες ε, στρεβλώσεις ε, των προηγούμενων νομοθεσιών που έχουν εγκρίνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που σήμερα δυναμητίζουν την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και μάλιστα είναι αντίθετα με τις αρχικές προθέσεις, δηλαδή το να καταστεί να είναι η οικονομική ένωση πιο σταθερή. Τώρα, όσον αφορά τις εργασίες για αυτήν την νομοθεσία, θα είναι μια νομοθεσία που έχουμε δύο βασικά προβλήματα. Το ένα είναι πιο μεγαλύτερο και είναι Θα πρέπει όμως να το ξεπεράσουμε γιατί διαφορετικά θα είμαστε βυθισμένοι στην αστάθεια του συστήματος όπως το βιώνουμε αυτές τις μέρες και το άλλο πρόβλημα είναι τεχνικής ε, φύσης γιατί ελπίζω πως εδώ θα έχουμε την ευκαιρία, όπως είπαμε και από την πρώτη αυτή συνάντηση, να κατανοήσουμε βαθύτερα πως τα σχέδια εγγύησης ε, καταθέσεων λειτουργούν, τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ε, λειτουργούν στα άλλα μέρη του κόσμου. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαφορετικό ζώο από τα υπόλοιπα. Έχουμε πολλές ιδιαιτερότητες, έχουμε θεσμούς ε, που είναι μοναδικοί στο είδος τους, στον κόσμο και αναφέρομαι κυρίως στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Άρα πρέπει να λάβουμε ε, υπόψη αυτές τις ιδιαιτερότητες. Ε, πρέπει λοιπόν να σταθεροποιήσουμε και να εξασφαλίσουμε τις εγγυήσεις ε, των καταθέσεων εντός των τραπεζών ε, της Τραπεζικής Ένωσης και πρέπει να πάμε πολύ πιο πέρα από την πρόταση και την προσέγγιση της Κομισιόν. Ένα σύστημα το οποίο βασίζεται καταρχάς ε, σε τρία βήματα πολύ αργό, το οποίο να ξεκινά να λειτουργεί το 2024 δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. 8 χρόνια ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Από την άποψη λοιπόν του χρονοδιαγράμματος δεν έχουμε όλο αυτό το χρόνο. Θα πρέπει να ξεκινήσει πιο γρήγορα, κάτι γνώμη μου. Τώρα, όσον αφορά τις ίδιες τις διατάξεις, και εδώ πιστεύω ότι για να δημιουργηθεί ένα σύστημα αξιόπιστο, το οποίο να ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη σταθεροποίησης του συστήματος, ένα σύστημα το οποίο θα χρηματοδοτείται βασικά από τις τράπεζες ε, δεν μπορεί να σταθεί γιατί παρουσιάζει πολλές ελλείψεις. Χρειάζεται υποστήριξη ισχυρών θεσμών όπως και στα άλλα μέρη του κόσμου. Στις ΙΠΑ, το σύστημα αγγίζης καταθέσεων στηρίζεται από μια γραμμή που πιστοτική που είναι αφιερωμένη σε αυτό από το, ε, Γενικό Ταμείο του Κράτους ε, και αντίστοιχα σε άλλες χώρες. Σε αυτά τα μοντέλα θα πρέπει να βασιστούμε. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εντός αυτού του συστήματος να παίζει ένα κύριο ρόλο. Διαφορετικά, οποιαδήποτε διάταξη που θα προβλέπει αποκλειστικά μια στήριξη αποκλειστική του ιδιωτικού τραπεζικού συστήματος με διαφορετικά είδη συμβολής επί τη βάση της διάστασης ή το κινδύνου δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει και σας δίνω ένα παράδειγμα της χώρας μου όπου το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων χρηματοδοτείται από τις συμβολές των τραπεζών. Σήμερα αν πάμε να δούμε την αναφορά του Ταμείου Προστασίας των Καταθέσεων, διαπιστώνει κανείς ότι στην Ιταλία υπάρχουν 5 δισεκατομμύρια καταθέσεις που έχουν δικαίωμα να καλύπτονται από αυτό το Ταμείο, αλλά αν δεν θυμάμαι καλά, ε, το Ταμείο αυτό έχει στη διάθεσή του πολύ λιγότερα δίση. Είναι δηλαδή τη τάξη των 7 δισεκατομμύριων οι υπάρχουσε εγγυήσει, ενώ οι καταθέσει ανέρχονται στα 550 δι. Αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα. θα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση που να σταθεροποιεί το σύστημα και όπως είπα εξ αρχή να μπορέσει να εξηγιάνει τις τρευλώσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος που εκκρεμούν λόγω ατελών νομοθεσιών που είχαν γίνει στο παρελθόν, ίσως λόγω της ε, όθησης, της βιασύνης ή της κρίσης. Πάντως είναι μια κατάσταση που πρέπει να εξηγιανθεί. Σας ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει Η αλήθεια είναι ότι το 7% για τα 500 δις είναι κάτι παραπάνω από 1%. Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε κυρία εισηγήτρια. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποια πράγματα γενικά, αν μου επιτρέπετε. Σε ό,τι αφορά το σύστημα αυτό. Είμαι αντίθετος για πολιτικούς και οικονομικούς ε, λόγους. Ε, από πολιτικό, μάλλον ε, να αναφερθώ γενικά σε ό,τι αφορά το πολιτικό και το οικονομικό. Δεν έχουμε πιστεί ότι τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να παραμείνουν ε, χρήσιμα για το κοινωνικό του σύστημα. Καλό ακούγεται αυτό στην θεωρία, αλλά ουσιαστικά είναι περαιτέρω μια Ένωση Μεταφορών, οι βόρειες τράπεζες προς βοήθεια των νότρων τραπεζών, οι οποίες είναι πολύ πιο ευάλωτες από τη Βόρεια Ευρώπη. Και τελικά επιβαρύνεται ο φορολογούμενος της Βόρειας Ευρώπης, άρα μεταφορά από Βόρεια σε Νότια Ευρώπη. Και η πολιτική της ΕΚΤ βασίζεται σε μια τέτοια αντίθεση. Δεν θέλω λοιπόν να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αυτά για το πολιτικό σκέλος, για το οικονομικό σκέλος τώρα. Από οικονομικής άποψης ε, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ακαδημαϊκές μελέτες τις οποίες θα τις ε, παρέχω, θα παρέχω στις επόμενες ε, συναντήσεις για το ότι ένα τέτοιο σύστημα υπονομεύει τη σταθερότητα των οικονομικών συστημάτων και άρα δεν ισχύουν όσα μα λένε οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι και το καθεξή ότι αυτό ε, σημαίνει μεγαλύτερη σταθερότητα και επίση αυτό αυξάνει τον ε, moral hazard, τον ηθικό κίνδυνο, τη συγκέντρωση κεφαλαίων και έχει αυξηθεί αυτή η συγκέντρωση κεφαλαίων στις μεγάλες τράπεζες, οι οποίες υπολογίζουν ότι εν πάση περιπτώσει θα παρέμβει το κράτος για την ε, ιδιωτικοποίηση του κέρδους και την ε, κοινωνικοποίηση, την αμοιβαιοποίηση των απολειών, των ζημιών. Κάποιοι θα μιλήσουν για ένα σύστημα με bail-in και ότι θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τις τράπεζες, αλλά όσοι έχουν λίγη κοινή λογική θα καταλάβουν ότι όταν κάτι πάει στραβά στις μεγάλες τράπεζες θα οι απώλειες είναι τόσο μεγάλες που τελικά οι φορολογούμενοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πληρώσουν την ύφη. Και 100.000 ευρώ ανά άτομο και αυτό είναι τελείω παράλογο γιατί πραγματικά αν συμβεί κάτι κανείς δεν θα μπορέσει να δώσει τόσο πολλά λεφτά και θα πιεστούμε ακόμα πιο πολύ από ό,τι σήμερα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά και να μπορούμε να δώσουμε τα 100.000 στον καθένα. Αυτό θα σημαίνει τεράστιο πληθωρισμό και μείωση της αξίας των χρημάτων και ξαφνικά θα γίνουν όλα αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά για το ποσό των 100.000, το οποίο ισχύει για πολλές χώρες, είναι τίποτα αυτό. Το χρυσό χάπι, αν θέλετε. και σε ό,τι αφορά τα πλούσια και φτωχά κράτη-μέλη. Προσβλέπω στις μελλοντικές συνεργασίες ε, με τους ε, συναδέλφους και θα ήθελα να σας πω ότι ε, πρόκειται να σας παρουσιάσω συγκεκριμένα επιχειρήματα, αλλά ήθελα ήδη από σήμερα να εκφράσω την αντίθεσή μου σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στο Catch the Eye. So, okay, we give Τρία λεπτά. Μπάλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Έστεντε Λάγκε για την ε, εξαιρετική εισαγωγή στο θέμα. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρόταση του Νοεμβρίου, πρέπει να σας πω ότι εμένα με εξέπληξε λίγο. Δεν την καταλαβαίνω τόσο την πρόταση. Βασιζόμαστε στην πρόταση της συνένα των Προέδρων που δεν έχει τύχη διαβούλευση, ούτε έχει νομιμοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να πω, επειδή είμαστε σε μια πρώιμη φάση της συζήτησης θα ήθελα κυρίως να θέσω ερωτήσεις. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τον νομοθέτη στον τριμερή διάλογο. Πώς ε, ορίσατε το έτος 2019 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς τοποθετείται για την ατζέντα, για την καλύτερη ρύθμιση, για το better regulation και σε ό,τι αφορά τις εξάντε μελέτες πριν από την νομοθετική πρόταση καθώς και τις θέμα των ε, διαβουλευσεών. Και σε ό,τι αφορά την ατζέντα του Better Regulation θα πρέπει να λεφθεί υπόψη εδώ στο έντις. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν με την πρόταση αυτή κανονισμού θέλει τώρα να τα θεωρηθεί κατεπηγόντως δεν θα πρέπει να κοιτάξει πιο κατεπηγόντων σε την εφαρμογή και τη συνεκτική εφαρμογή ήδη ψηφισμένων νομοθεσιών, νομοθετημάτων. Γιατί πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει τα νομοθετημάτα τα σχετικά και δεν θα έπρεπε να φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εθνικά συστήματα να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο, στις περιπτώσεις moral hazard, δυτικού κινδύνου και δεν θα ήταν πιο κατεπήγον να κοιτάξει την εφαρμογή της αρχής του bail-in με 8% ελάχιστο και την ίση αντιμετώπιση των πιστωτών. Και επίσης αναρωτιέμαι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανησυχεί γιατί κάποια κατημέλη προωθούν το έντις και κάποια άλλα το αποφεύγουν. Πόσο συνδυάζονται αυτά και πώς ε, ε, λαμβάνει υπόψη τους ισολογισμούς των τραπεζών και πως λαμβάνει υπόψη είναι το γεγονός ότι πολλές τραπέζες έχουν υπερβολικές επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα όπου τα κράτη είναι ακόμα υπερχρεωμένα. Δεν θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει πιο πολύ το θέμα της μείωσης ε, του κινδύνου. Πιο πολλές ερωτήσεις έχω παρά απαντήσεις. Όποιος μιλάει για μείωση, ε, μάλλον για την ε, Τραπεζική Ένωση, θα πρέπει να κοιτάξουμε βασικά την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να επανέλθουμε στην αρχή ευθύνη για τον κίνδυνο και θα πρέπει να μειωθούν περτέρω οι κίνδυνοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αποφάσισε και δεσμεύτηκε πέρα από την πρόταση έντης να προτείνει και μέσα για την μείωση του κινδύνου όχι, όποιος έχει προχωρήσει τόσο πολύ σε ό,τι αφορά με το ΕΔΙΣ, ε, σίγουρα θα μπορέσει μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει σχετικές προτάσεις. Ευχαριστώ. Πολλά θέματα ακούσαμε ήδη και γι' αυτό λοιπόν θα προσπαθήσω να είμαι σχετικά σύντομος. Καταρχάς, μου προκαλεί έκπληξη το γεγονό ότι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν χρειάστηκε μελέτη αντικτύπου γιατί το 2010 έκανε ήδη μια μελέτη αντικτύπου. Εγώ κοιτώντα ε, το ημερολόγιο διαπιστώνω ότι το 2016 έχουμε φτάσει πλέον. Τα τελευταία 6 χρόνια νομίζω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα τα οποία προφανώς θα πρέπει να αποτυπωθούν σε μια νέα μελέτη αντικτύπου. Πού να ληφθούν υπόψη το 2010, πόσο μάλλον όλες οι λεπτομερείς προτάσεις του ΙΔΙΣ. Δεύτερο θέμα. Edis. Το E είναι από το insurance. Από τη, τη μεταβατική όμως λύση για τη μακροπρόθεσμα. Δεν θα πρέπει να είναι μόνο ένα σύστημα ασφάλειας, αλλά ένα σύστημα εγγύσεων, ένα ενιαίο σύστημα Και θεωρώ ότι ακόμα και ο όρος είναι εσφαλμένος, ο όρος τον οποίο επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της και για πολλές, σε πολλές ανακοινώσεις τύπου μιλάει για τις ασφάλειες αυτές, αλλά για λόγους ε, πληρότητα θέλω να πω ότι αυτό προκαλεί ερωτήματα. Επόμενο θέμα. Αν θέλουμε να υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα, αναρωτιέμαι γιατί δεν έχουμε δημιουργήσει ίσους όρου συνταγωνισμού. Γιατί κάνουμε διάκριση μεταξύ αυτών που είναι μέσα στο ευρώ και αυτού που δεν είναι ακόμα μέσα στο ευρώ και αυτού που ποτέ δεν θα μπουν στο ευρώ. Οι οποίοι στα εθνικά του συστήματα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ 0, 0,5%, 0,8%. Ενώ μέσα στο ευρώ μόνο το 0,8% μπορούμε να ε, επιλέξουμε. Είναι αυτό θεωρή δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό μακροπρόθεσμα, θα δημιουργήσει στραβλόψεις Μαζικέ. Και γι' αυτό λέω με πάσα σαφήνεια σε ό,τι αφορά τη ΣΥΠΑ. Εδώ πέρα δεν υπάρχει επιρροή. Δεν ανακύπτουν τα θέματα αυτά. Επόμενο θέμα. Αν θέλουμε να το θέσουμε αυτό σε όλα τα επίπεδα για όλε τι τράπεζε, θα πρέπει να κοιτάξουμε και το ερώτημα κατά πόσον ε, θέλουμε και πρέπει να κάνουμε ε, μελέτη ποιότητας ε, των στοιχείων, των περισσοκών στοιχείων, να δούμε τι σημαίνει σε όλες τις τράπεζες που βρίσκονται υπό την εποπτεία των, ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 8.000 τράπεζε, δεν ξέρω πόσε είναι. Θέλουμε πραγματικά να το κάνουμε αυτό. Και ένα άλλο θέμα το οποίο θα συζητήσω αύριο με την Επιτροπή Φριστά και το θέμα τη πρόληψη και σε ό,τι αφορά την εξυγίανση. Μήπως σε τελική ανάλυση έχουμε μόνο το θέμα της ε, εξυγίανσης, της εκαθάρισης. Ε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έχω πάρα πάρα πολλά ερωτήματα, όπως πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Θέλουμε μεγαλύτερη σαφήνεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην παρούσα φάση όμως θέλω να πω ότι το τρέχον νομικό πλαίσιο θεωρώ ότι επαρκεί αν και εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε να φροντίσει ότι όλα τα κρατημέλη θα εφήρμοζαν αυτό το πλαίσιο στις εθνική νομοθεσία. Θεωρώ ότι αυτό φτάνει και περισσεύει. Thank you, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε είναι σαφές ότι στα πλαίσια αυτής της ανταλλαγής απόψεων ακούει κανείς τα πάντα γύρω από τις προτάσεις αυτής της μορφής ασφάλισης των καταθέσεων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω καταρχάς ότι το χρονοδιάγραμμα το οποίο μας προτείνεται έτσι ώστε να υπάρξει σταδιακή εφαρμογή είναι κάτι που πρέπει να επιταχυνθεί γιατί η Τραπεζική Ένωση αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα βλέπουμε την αστάθεια η οποία επικρατεί και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το μοντέλο αυτό το ταχύτερο δυνατόν με υψηλότερη ταχύτητα. Θα ήθελα να θέσω και εγώ κάποια από τα θέματα τα οποία ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έθεσαν πολλοί συνάδελφοι. Λοιπόν, την ανάγκη αναθεώρησης της, του καθεστώτος του νομικού, του δημοσίου χρέους ως αντικειμένου ελευθέρου από κίνδυνο. Και στα πλαίσια της Βασιλείας είναι αβέβαιο για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα και υπάρχουν τράπεζες στο εσωτερικό ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που περιλαμβάνουν τμήμα του δημοσίου χρέους στο εσωτερικό της αγοράς. Νομίζω ότι στα πλαίσια λοιπόν της κοινή αυτής αγοράς κεφαλαίων θα πρέπει να μην υπάρχουν διακρίσεις και αυτό θα βελτιώσει γενικά την αποτελεσματικότητα της ζώνης ευρώ. Τώρα σχετικά με τα ανώτατα όρια των τμήματων που ε, γίνονται αντικείμενο εγγύησης, θυμίζω ότι δύο χώρες έχουν, ε, έχουν υποστεί τέτοιου είδους καταστάσεις όπως η Ελλάδα και το θέμα είναι βέβαια ποια είναι τα οικονομετρικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί και το δημόσιο χρέος σαν τμήμα του προβλήματος. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για να σταθεροποιηθεί το χρηματοπιστωτικό πρέπει να υπάρξει υψηλότερο επίπεδο εποπτείας και στα πλαίσια του, ενός του πυλώνα της Βασιλείας. Θα πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια των ε, στοιχείων ε, που περιλαμβάνονται στον πυλώνα της Βασιλείας και νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε πιο βέβαιοι και σίγουροι και σε σχέση με τα σύμφωνα σταθερότητας και για τον σημαντικό ρόλο τον οποίο έχουν να παίξουν οι τράπεζες ε, γενικότερα στο θέμα της ε, πολιτικής, της οικονομικής αλλά και της δημοσιονομικής. Νομίζω ότι ε, δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα τη διαδικασία εγγύησης και διασφάλισης των καταθέσεων. Υπάρχουν αμφιβολίες και σε σχέση με τον ρόλο και τον χαρακτήρα λοιπόν του δημοσίου χρέους ε, και νομίζω ότι είναι ευθύνη όλων μας να βρούμε κάποιες λύσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους οι οποίοι μίλησαν. Είναι σαφές ότι υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις όμως τις οποίες θα πρέπει να θέσω κι εγώ. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει ε, χαρακτηριστικά πολεμικά σε εισαγωγικά θα έλεγα έντονης αντιπαράθεσης. Είναι απαραίτητο όμως η συζήτηση να γίνει. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην δημιουργία, στην ε, ολοκλήρωση των πυλώνων αυτών απαιτείται τεράστια προσπάθεια και η προσπάθεια αυτή δυστυχώς δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου εύκολη. Τώρα σε σχέση με την αμοιβεοποίηση των κινδύνων δεν είναι θεωρητικό το θέμα. Το θέμα αυτό είναι όμως ε, κάτι το οποίο δημιουργεί αντιθέσεις σε πάρα πολλά κράτη-μέλη και είναι σαφές ότι δεν μπορεί να προχωρήσουμε σε δυνατότητες αμοιβεοποίησης αν δεν υπάρχουν αντισταθμήματα. Δεν μπορούμε επίσης να αντιστοιχίσουμε τα πάντα με τα πάντα, δεν είναι δυνατόν. Γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται να σημειώσουμε κανένα βήμα προόδου. Νομίζω όμως ότι βρισκόμαστε σε καλά χέρια και ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί με επικοδομητικό τρόπο. Excellent. Ο κύριος Μαυρίδης. Thank you, Chairman. I think that, um, Πιστεύω ότι η συζήτηση που κάνουμε είναι κάτι παραπάνω από ότι ένα απλό σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Δεν θα λύσουμε τις τεχνικές στοιχείες, ούτε θα τις συζητήσουμε εκτεταμένα σήμερα. Είναι η πρώτη συζήτηση. Νομίζω όμως πως η συζήτηση αυτή σε σχέση με το σύστημα εγγύησης καταθέσεων και την Τραπεζική Ένωση έχει να κάνει με περισσότερα από ό,τι απλά η Τραπεζική Ένωση. Εγώ κατανοώ ότι βρισκόμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε κοινού κανόνες. Όμως αυτοί οι κοινοί κανόνες θα πρέπει να είναι και αμερόληπτοι. Και πιστεύω πως μια τραπεζική ένωση χωρίς ένα τρίτο πυλώνα δεν είναι απλά ατελής, είναι σίγουρα και πολύ μεροληπτική. Και θα σας δώσω και κάποια παραδείγματα. κάποιες απαντήσεις που καθιστούν σαφές ότι είναι μεροληπτική μια τέτοια κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν απόλυτα σαφής για αυτό το θέμα. Χωρίς ένα τρίτο πυλώνα, βασικά η Τραπεζική Ένωση είναι ε, ε, ε, είναι, ε, μάλλον συμπεριφέρεται διαφορετικά απέναντι στους καταθέτες γιατί δεν τους μεταχειρίζεται όλους με τον ίδιο τρόπο. Είναι έμεσα δε ε, άνηση και προς την Τραπεζική Ένωση γιατί δεν μεταχειριζόμαστε, δεν αντιμετωπίζουμε τις τράπεζες τις ιδιωτικές με τον ίδιο τρόπο, δεν έχουμε ισότιμο πεδίο που να μπορούν να ανταγωνιστούν και σας δώσω ένα πολύ καλό παράδειγμα. Μια ιδιωτική τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια πρέπει να ανταγωνιστεί με μια τράπεζα κάπου στη Γερμανία όπου οι δύο τράπεζες ε, είναι εγγυημένες από διαφορετικές κυβερνήσεις. Και φυσικά αυτό έμεσα δημιουργεί ανταγωνιστικό πλονέκτημα. Δύο λόγια ακόμα. Θυμούμε ότι όταν είχαμε τον διορισμό των επιτρόπων πριν από 1,5 χρόνο, η συζήτηση τότε δεν ήταν αν θα εφαρμοστεί ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων, αλλά ε, το θέμα ήταν το πότε. Τώρα φαίνεται ότι ορισμένοι έχουν αλλάξει γνώμη. Τώρα, όσον αφορά το FTIC, βεβαίως αναγνωρίζουμε τις διαφορές, αλλά η συζήτηση με το FTIC ποτέ δεν ήταν να το καταργήσουμε, αλλά να το, να το επεκτείνουμε και μάλιστα να αυξηθεί το μάξιμο ποσό. Ένα ερώτημα το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι είναι απόλυτα θεμητό είναι το θέμα του ηθικού κινδύνου που είναι πολύ, πολύ θεμητό ζήτημα, επαναλαμβάνω. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έγινε ε, ο πρώτος και δεύτερος πυλώνας και μετά ο τρίτος, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το θέμα του ηθικού κινδύνου. Αν κάποιο αναζητεί τραπεζική ένωση με ένα σύστημα αγγίσης καταθέσεων χωρί ηθικό κίνδυνο, τόσο αυτός ο άνθρωπο δεν επιθυμεί την ύπαρξη του σχεδίου εγγύηση καταθέσεων. Γιατί ο ηθικός κίνδυνο ή ένας περιορισμένος ε, ποσοστό, εν πάση περιπτώσει, τέτοιου κίνδυνου θα υπάρχει πάντοτε και πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ήταν ο Ευχαριστώ, Ρίτσαρντ. Ε, ευχαριστώ. Όταν ε, ρώτησε η λίδα γιατί, υπάρχει τύπης η δέσμευση των 100 μελών να ολοκληρώσουν την Τραπεζική Ένωση, αλλά υπάρχει και ε, μια λογική πίσω από όλο αυτό, διότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων στο επίπεδο όπου κανείς εποπτεύει τις τράπεζες και τον κίνδυνο σε αυτές, αυτές που είναι υπό την εποπτείωση. Είναι προφανής η εξήγηση του γιατί, αλλά υπάρχει πάντοτε και η εμπειρία της κρίσης που δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη αντασφάλισης των εθνικών συστημάτων εγγύησης καταθέσεων έναντι μεγάλων συστημικών γεγονότων που μπορεί να ξεπεράσουν την δυνατότητα απορρόφησης ζημιών της εθνικής αρχής και πιστεύω ότι γι' αυτό τα εθνικά συστήματα εγγύηση καταθέσεων μπορεί να φανούν αφαιρέγγια και το ξέρουμε αυτό από την εμπειρία μας και γι' αυτό και η εξασφάλιση εγγύηση έναντι των συστημικών σοκ είναι ε, μια εγγύηση για τη σταθερότητα του συστήματος. Τώρα, όταν μιλάμε για διασυνοριακές τράπεζες με θηγατρικές, βλέπουμε ότι οι θηγατρικές συμβάλλουν στα εθνικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων του εις χώρας υποδοχής. Οπότε, αν μια μεγάλη διακρατική τράπεζα πτωχεύσει και έχει θυγατρικές σε μια άλλη χώρα, τότε η Εθνική Αρχή θα πρέπει να καλύψει. Υπάρχει ήδη δηλαδή μοιρασιά του βάρους όσον αφορά τις διακρατικές τράπεζες. Κάτι ακόμα που θέλω να παρατηρήσω για αυτή τη δύσκολη σχέση ανάμεσα στο ημείωση κινδύνου και στη μοιρασιά την αμοιβιοποίηση του κινδύνου γιατί πιστεύω πως είναι πολύ περίπλοκο θέμα και δεν μπορούμε απλά να λέμε ότι πρώτα μπορούμε να μειώσουμε στο μηδέν το κίνδυνο να, μειώ, να, να το κίνδυνο και έπειτα να οικοδομήσουμε το μηχανισμό αμοιβιοποίησης του κινδύνου. Και εγώ ήδη εκπλήσωμαι, αλλά νομίζω ότι τα όσα είπε ο Φίλιπ Λάμπερτ ήταν λογικά. Νομίζω λοιπόν πως πρέπει να εξετάσουμε αυτούς τους δύο μηχανισμούς ε, παράλληλα. Θα πρέπει δηλαδή να φτιάξουμε ταυτόχρονα και τον μηχανισμό μείωσης του κινδύνου και τον μηχανισμό μοιρασιάς του κινδύνου. Σας ευχαριστώ. Νότης Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχαμε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων, διότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ε, ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να προστατεύσει πραγματικά τους καταθέτες σε περίπτωση πτώχευσης των τραπεζών, να έχουν τη δυνατότητα οι καταθέτες να αποζημιωθούν μέχρι ένα καθορισμένο όριο βέβαια και έτσι να αποκατασταθεί η σταθερότητα στην ίδια τη χρηματοπιστωτική αγορά. Βεβαίως το ερώτημα μπαίνει ότι ε, πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να αποφεύγονται οι πτωχεύσεις των τραπεζών που αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ένα ενισχυμένο σύστημα εποπτείας και πολύ περισσότερο σε τράπεζες οι οποίες ε, έχουν προβληματικούς ισολογισμούς, τράπεζες οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε παράγωγα, σε επισφαλή ομόλογα και έχουμε δει το πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει ήδη με την Deutsche Bank. Το επόμενο θέμα βεβαίως αφορά την ίδια την Ελλάδα, διότι στην Ελλάδα προκειμένου να υπάρξει αυτή η εγγύηση ουσιαστικά των καταθέσεων, να υπάρξει η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, επιβλήθηκε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών η οποία βεβαίως συνδυάστηκε με πάρα πολύ σκληρά μέτρα. Συνδυάστηκε με μνημόνια, συνδυάστηκε με μέτρα τα οποία έχουν μειώσει τους μισθούς, τις συντάξεις, έχουν κοινωνικοποιήσει τις ζημιές, δηλαδή έχουν περάσει όλες οι ζημιές ε, ουσιαστικά εις βάρος των ίδιων των φορολογουμένων και του ελληνικού λαού. Και μιλώντας για τα σκληρά μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί, αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει ως πρόβλημα σημαντικότατο στην Ελλάδα και το οποίο ανέδειξα σε αυτή την, ε, στη συνεδρία που κάναμε με τον κύριο Ντάισεμπλουμ είναι τα κόκκινα δάνεια τα οποία υπάρχουν. Τα κόκκινα δάνεια τα οποία με το τρίτο μνημόνιο, με την έγκριση της Τρόικας, την επιβολή μάλλον της γνώμης της Τρόικας και του Eurogroup, στο οποίο προείσταται ο κύριος Ντάισεμπλουμ, ε, πάνε για να πουληθούν, να πουληθούν στα funds, να πουληθούν στα κοράκια. Και τον ρώτησα γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε την λύση της Ιταλίας. Μια λύση την οποία σε αυτήν εδώ την αίθουσα στήριξε και ο κύριος Ντράγκη. Δηλαδή τα κόκκινα δάνεια, όπως συμβαίνει στην Ιταλία, να μπορούν υπό μορφή ABS να δοθούν ως εγγύηση, ως collaterals από τις Ιταλικές τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό ήταν ένα ερώτημα το οποίο έθεσα στον κύριο Ντάισεμπλουμ. Νύπτητα σχήρα στους πόντιο Πιλάτο, δεν απήντησε. Περιμένω βέβαια την απάντηση του κυρίου Δράγκη σε ερώτηση που κάναμε. Διότι το θέμα είναι να υπάρξει ίση μεταχείριση και των δανειοληπτών και στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Και αφού πράγματι έχει βρεθεί μια λύση που δρομολογείται στην Ιταλία, την οποία αποδέχεται και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με του όρου που μα εξήγησε εδώ ο κύριο Δράγκη νομίζω ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί να υπάρξει η ίδια απάντηση στο θέμα αυτό και για τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα προκειμένου οι δανειολήπτες να μην χάσουν τα σπίτια τους. Επομένως κύριε Πρόεδρε κλείνοντας νομίζω ότι είναι πολλά τα ζητήματα που είναι ανοιχτά. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να συζητήσουμε και άλλες λεπτομέρειες στις, στα επόμενα στάδια των συζητήσεων. Πάντως πιστεύω ότι η συζήτηση θα είναι ενδιαφέρουσα αλλά πρέπει επιτέλους να ληφθούν σοβαρά μέτρα για ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ja, Dank, äh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Όντως, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη συνένεση για το ότι όλα θέλουμε να τα κάνουμε για να πετύχουμε τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη. Ωστόσο, αναρωτιέμαι στην παρούσα φάση κατά πόσον τα μέτρα αυτά τα οποία συζητούμε σήμερα σε ό,τι αφορά την ε, αμοιβεοποίηση των εγγύησεων πραγματικά είναι το σωστό και ενδεικμένο μέσο. Το θέμα της αιτίας της αστάθειας των τραπεζών. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν για το θέμα αυτό. Και έτσι νομίζω ότι γρήγορα καταλήγουμε στο μεγάλο πρόβλημα ότι οι τράπεζες ε, έχουν επιβαρυνθεί με κρατικά ομόλογα και γι' αυτό δεν μπορούν λοιπόν να αντιδράσουν με αμοιβαιοποίηση. Θα έπρεπε να δοθεί συντελεστή ρίσκου στα κρατικά ομόλογα και αυτό συζητήθηκε στην Τραπεζική Ένωση. Και αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί η Κομισιόν δεν έκανε πρωτα... την πρόταση αυτή ακριβώ. Σε ό,τι αφορά και τη μείωση του χρέου των κρατών, πώ μπορούμε να μειώσουμε τα ελλείμματα. Ούτε αυτό είναι στο επίκεντρο. Αυτό που είναι στο επίκεντρο είναι η αμοιβαιοποίηση της ευθύνη σε ό,τι αφορά τις, ε, την ασφάλεια των καταθέσεων. Ετέθησε πάρα πολύ γρήγορα στην ημερήσια διάταξη χωρίς να αποκαλυφθούν οι πραγματικοί λόγοι. Είναι σχεδόν πανικόβλητη ανταπόκριση, αντίδραση. Το θέμα λοιπόν είναι τι έχει γίνει με τις αποφάσεις που ήδη έχουν ληφθεί, έχουν εφαρμοστεί οι αποφάσεις αυτές γιατί σε κάποιε χώρε δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα ακούμε. Γιατί να κάνουμε το δεύτερο βήμα, αν δεν έχει γίνει καν το πρώτο. σε ό,τι αφορά τα εθνικά ταμεία ασφαλίσεων. Θέλω να μα απαντήσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ερώτηση αυτή. Ιδάλλως δεν έχει νόημα να κάνουμε καινούργια νομοθεσία και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια πιο σωστή ανάλυση μιλώντας με τους ειδικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας λένε ότι α, βέβαια, αλλά το πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα δεν υπάρχει στις αποκεντρωμένες ε, περιοχές. Μα τότε το θέμα δεν είναι η ασφάλεια των καταθέσεων. Το θέμα είναι πώ θα πετύχουμε τη ρευστότητα σε κάποια τμήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ τίθεται το θέμα του κατά πόσον ε, δίνουμε τη σωστή λύση στο πρόβλημά μα. Τελευταίο θέμα το οποίο θέλω να θίξω. Σήμερα το πρωί είχαν την τιμή ως ε, αντιπρόεδρος της ε, Intergroup για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να παρουσιάσω μια μελέτη για το θέμα του κόστους ρύθμισης για τις μικρομεσαίες τράπεζες. Είχαμε κάποια εμπειρικά στοιχεία ήδη τότε σχετικά με την νομοθεσία που ψηφίσαμε και το πώς έχει αντικτύπωση στις τράπεζα ανάλογα με το μέγεθός του. Ο συνάδελφος Φέρμπερ έθεσε το θέμα του ανταγωνισμού και του ίσου ανταγωνισμού. Εγώ θεωρώ πριν αρχίσουμε να κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις για την αμοιβαιοποίηση τη ε, ευθύνη θα πρέπει να λύσουμε επακριβώς ποιε θα είναι οι συνέπειε στον ανταγωνισμό. Και να δώσω και ένα παράδειγμα. Εσφαλμένα διατείνεται πάρα πολλοί κόσμο ότι... Στη... Ναι, συγγνώμη λέει ο πρόεδρο, δεν έχετε άλλο χρόνο. Ναι, λυπάμαι, λέει ο πρόεδρο. Μάλιστα, δεν, ε, δεν έχουμε υπερβολικά πολλές τράπεζες, αλλά η κατάσταση έχει να κάνει με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και είναι συγγνώμη πρόεδρε, το θέμα είναι τι ε, γίνεται και με τον ανταγωνισμό. Αυτό ήθελα να δείξω. Ευχαριστώ πολύ ο Πέτρος Εισαγωγικά θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπε στην αρχή ο προηγούμενος ομιλητής. Έχουμε λοιπόν ένα στόχο. Θέλουμε να ενισχύσουμε την Τραπεζική Ένωση. Το θέμα είναι το πώς θα το πετύχουμε αυτό. Αυτό. Σε αυτό αποκλίνουν οι απόψει. Α σκεφτούμε λοιπόν κάποιε βασικέ αρχές για την ενίσχυση τη Τραπεζικής Ένωση. Αυτό που είναι σαφέ, πιστεύω είναι ότι δεν μπορούμε να επαναχωρήσουμε σε αυτά που έχουμε ήδη πετύχει. Αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο λειτουργίας για την προστασία των καταθέσεων, όπως και με τη σταθερότητα σε απόλυτους αριθμούς σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργία. Όπως έχει η σημερινή νομοθεσία, έχουμε δημιουργήσει κάτι το οποίο ως τώρα το αναζητούσαμε στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει λοιπόν μόνο ασφάλεια των καταθέσεων μέσω ενός paybox και έχουμε και ε, εναλλακτική και την εκαθάριση Υπάρχει και κάτι στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που δεν υπήρχε ω τότε. Είχε βοηθήσει πάρα πολύ σε διάφορες περιστάσεις. Το μέτρα Early Intervention με χρηματοδότηση από πλευρά των ε, τραπεζών, όχι από τρίτους, που αποτρέπουν παρέμβαση του φορολογούμενου και του, ταμείου, του Εθνικού Ταμείου Ασφάλειας Καταθέσεων. Το εργαλείο λοιπόν αυτό να μην το αφήσουμε κατά μέρος να προστατεύσουμε την εργαλειοθήκη και να μην την περιορίσουμε. Και έτσι να προωθήσουμε την χρήση της χρηματοδότησης. Επίσης όμως θα πρέπει να επιδιώξουμε το στόχο μας και στις χώρες όπου δεν υπάρχουν τόσα πολλά εργαλεία για την προστασία των καταθέσεων ακόμη. Και δεν γίνονται αντιληπτά τα μέσα αυτά από τον κόσμο. Να ενισχυθούν τα μέσα αυτά, χωρίς όμως να καταστραφούν τα συστήματα και να στρεβλωθούν τα συστήματα της χώρας και να μειωθεί και η εμπιστοσύνη στα συστήματα αυτά. Δεν θα είναι θετικό αυτό για κανέναν αν στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, σταθερά κράτη καταλήξουν στο τέλος να βρίσκονται σε πιο δύναμη κατάσταση από ότι στην αρχή της διαδικασία. Αυτό να το προσέξουμε σε κάθε περίπτωση και ως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσέξουμε το, εστί, το εξής. Να μην μας συμβεί το εξής. Αυτό που έγινε για την με την νομοθεσία για την εκαθάριση. Πολλά μεταφέρθηκαν σε επίπεδο 2 και ως Κοινοβούλιο ασκήσαμε μαζική κριτική σε ό,τι αφορά το συντελεστή κινδύνου των παραγόντων ότι δεν, ήταν, δεν είχε διαμορφωθεί με τρόπο, τον τρόπο που είχαμε φανταστεί. Και να δούμε τι γίνεται με την ε, τρέχουσα πρόταση νομοθεσία. Όλα συνολικά μεταφέρονται σε επίπεδο 2 και ω κοινοβούλιο αντιμετωπίζουμε ακριβώ την ίδια κατάσταση όπω και τότε. Νόμιζα λοιπόν ότι κάτι θα είχαμε διδαχθεί από το παρελθόν και ένα από τα βασικά, από, μία από τις βασικές αξιώσεις θα πρέπει να είναι όλα αυτά τα θέματα να ληφθούν υπόψη και όλα αυτά να περάσουν σε επίπεδο 1, σε επίπεδο νομοθεσίας όπου εμείς θα είμαστε συνομοθέτες. Thank you. Ευχαριστώ. Κάποιες ερωτήσεις ε, απευθύνθηκαν προς την Κομισιόν. Είναι εδώ ο Πάτρικ Φέρσον. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομο. Μετά από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή, έχω τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι είναι σωστό η σημερινή οδηγία απαιτεί από την Κομισιόν να αναθεωρήσει την οδηγία και να προβεί στις απαραίτητες νομοθετικές προτάσεις μέχρι το 2019, το αργότερο, εμείς αποφασίσαμε να μην περιμένουμε μέχρι το 2019. Η πρόταση της Κομισιόν αφορά τον χαμένο τρίτο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης. Έχουμε δηλαδή έναν επόπτη Έχουμε ένα νέο ε, μηχανισμό εξυγίανσης ε, που αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά δεν έχουμε ένα νέο σύστημα εγγύησης καταθέσεων για τους πολίτες μας όταν ε, μια τράπεζα πεθάνει. Έτσι λοιπόν η αρνητική ανάμεσα στα κράτη και τις τράπεζες εξεκολουθεί να υπάρχει. Πιστεύουμε ότι το τραπεζικό σύστημα έτσι θα γίνει πιο αξιόπιστο, πιο ασφαλές και θα αυξηθεί και η εμπιστοσύνη των πολιτών. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ακούσαμε πάρα πολύ προσεκτικά αυτή την εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων. Πολλές θετικές παρατηρήσεις έγιναν και πρέπει να λάβουμε υπόψη το κόστος για το τραπεζικό τομέα. Οφείλουμε να αναδιερωτηθούμε πώς μπορούν οι συμβολές αυτές να αξιοποιηθούν χρειάζεται να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια για όλα αυτά και διαφάνεια. Επίσης πρέπει να εξετάσουμε τα θέματα ηθικού κινδύνου. Η πρόταση περιλαμβάνει ασφαλιστικές δικλείδες κατά της κατάχρησης του συστήματος, απαιτείται η εφαρμογή της ισχύουσας οδηγίας και η τελευταία πληροφορία που έλαβε η Κομισιόν είναι ότι έξι κράτη-μέλη θα έπρεπε να έχουν μεταφέρει φέρει αυτή την οδηγία φέτος την Άνοιξη. Πρέπει να δούμε και θέματα κληρονο... Ε, κληρονομιάς. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα συστήματα τα θεσμικά για την ασφάλιση των καταθέσεων που υπάρχουν σε κάποια κατημέλη να πρέπει να, συνεχίσουν την πολύτιμή του συμβολή στη σταθερότητα στα εν λόγω κρατημέλη. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα στην πρότασή μας. Ελπίζουμε ότι η μακροπρόθεσμη εφαρμογή 2024 επίσης θα συμβάλλει σε αυτό. Τρίτη μου παρατήρηση είναι ότι η Κομισιόν συμφωνεί απόλυτα με αυτού που είπαν ότι πρόκειται για αμοιβαιότητα των αμοιβαιοποίηση μάλλον του κινδύνου η Κομισιόν συμφωνεί ότι αυτά τα μέτρα θα πρέπει να συνοδεύονται και από μέτρα μείωσης του κινδύνου. Η ανακοίνωση της Κομισιόν υιοθετήθηκε μαζί με αυτή την πρόταση και δείχνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο. Έχουμε τις τα options, τα TILAC, την αφεργιότητα, το κίνδυνο των κρατικών χρεών, κρατικού χρέους κτλ. Προχωράμε λοιπόν φιλόδοξα το Συμβούλιο, οπότε κατάλαβα να ζητούν να έχουν κοινή θέση τον Ιούνιο, μια γενική κοινή θέση τον Ιούνιο. Εμείς προσβλέπουμε στην επικοδομητική συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Thank you. Και εγώ σας ευχαριστώ. Υποθέτω πως ε, η Κομισιόν με το Συμβούλιο δεν ε, τακώνονται για το δικαίωμα πρωτοβουλίας ε, της Κομισιόν η εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το χρονοδιάγραμμά μας τώρα. Νομίζω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες εκτός μίας συμφωνούν Νομίζω είναι μια καλή ισορροπία ανάμεσα στο να πάμε αργά και προσεκτικά και από την άλλη να μην χάσουμε χρόνο. Έγιναν πάρα πολλές και πολύ σημαντικές παρατηρήσεις. Ε, αν πάει κανείς λίγο προς τα πίσω, μετά από αυτά που ακούσαμε, θεωρείται, θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει ασφάλιση των εγγύησεων. Αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο πολίτης, ο μέσος πολίτης θέλει να υπάρχουν εγγυήσει ε, για, τα, για τις καταθέσεις του. Υπάρχουν εθνικά σχήματα τα οποία δεν το κάνουν αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να δίνουμε την εικόνα και την εντύπωση ότι δεν υπάρχει κανένα. Ε, και με μια απλή ενίσχυση ρευστότητα θα λυθούν όλα τα θέματα. Πολλοί συνάδελφοι λοιπόν μας είπαν ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε τα μέσα με τα οποία θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανησυχίες των πολιτών. Και γι' αυτό ακριβώς η πρόταση αυτή είναι μια αξιόλογη προς την κατεύθυνση αυτή πρόταση. Αυτό που είναι σημαντικό επίσης είναι και η παρατήρηση πολλών συναδέλφων ότι κάθε χώρα και κάθε εθνικό σχήμα προστασίας θα πρέπει να βγει ενισχυμένο. Αυτό το οποίο θα ήθελα να, για το οποίο θα ήθελα να προειδοποιήσω είναι η σύγκριση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε όμως δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε ένα οικοδόμημα εθνικών επιπέδων και γι' αυτό δημιουργούμε το ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αν εμείς βλέπουμε ε, τη δυνατότητα αυτή σαν μια μεταφορά από το εθνικό επίπεδο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε θα αποτύχουμε. Το θέμα είναι ότι η ευθύνη θα πρέπει να αναλυθεί σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Αν ακολουθήσουμε τη λογική αυτή του αποκλεισμού, τότε το σύστημα δεν θα δουλέψει. Σχετικά με την ανάμειξη, πολλές ομάδες αναφέρθηκαν στα προβλήμα, στο πρόβλημα αυτό και άκουσα εγώ κάποια στοιχεία όπως ας πούμε ε, τα θέλματα ρευστότητας. Um, discrepancy between uh, όπως επίσης και τα θέματα της φερεγγιότητας των πιστοτικών ιδρυμάτων και τις νομικές ρυθμίσεις που τα διέπουν. Άκουσα επίσης από διάφορες πλευρές και το θέμα του δημόσιου χρέους, όπως επίσης και κάποια στοιχεία τα οποία γενικά ελείπουν από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τώρα τουλάχιστον. Ε, εγώ και η Ντανούτα είχαμε μια κοινή εμπειρία. Ε, είπες ότι εξεπλάγεις γιατί συμφώνησες με τον Λάμπερτς, είπε η Ντανούτα. Ε, μου κάνει εντύπωση που συμφωνώ με τον Φίλιπ Λάμπερτς. Μα φυσικά και εγώ, και εγώ συμφωνώ με πολλά από τα στοιχεία τα οποία ανέφερε ο Λάμπερτς. Ένα είναι το πώς μπορούμε να συνδέσουμε νομικά το θέμα της μείωσης του κινδύνου με το θέμα της κατανομής του κινδύνου. Όπως επίσης ε, και το θέμα της στάθμισης του κινδύνου σε σχέση με την συνεισφορά προς το Ταμείο. Και θα πω επίσης προς τον κύριο Φέρμπερ ε, ότι υπάρχει το θέμα των μέσα, των έξω και των ίσως. Υπάρχουν ε, ε, εδώ κάποια σημεία τα οποία τίθενται και σε εθνικό επίπεδο και σε κοινοτικό επίπεδο και ακόμα δεν έχουν ε, διευκρινιστεί και για τον Πέτερ Σίμων θα ήθελα να ευχαριστήσω γιατί έχει συμπειρία στα θέματα αυτά σχετικά με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και σε σχέση με τον κίνδυνο ο οποίος είναι ενταγμένος μέσα στις νομικές ισχύουσες ρυθμίσεις και η προειδοποίησή σου για τη μη επανάληψη των λαθών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφύγουμε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν προς την καλή ελπίζω κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σεβαστήκαμε και τα χρονικά όρια γενικότερα. Το θέμα αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα και άκουσα πολύ σημαντικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Πολλά θα ήθελα να τα συζητήσω, αλλά θα τα κάνουμε σε διμερή βάση. το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς ε, τη μείωση των κινδύνων μέσω αύξησης του κεφαλαίου και όχι ε, μέσω της μείωσης των προϋποθέσεων ε, για, την, για τα θέματα της συνολικότερης πτώχευσης. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Νομίζω ότι στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει, ε, υπάρξει μια περίπτωση ε, πτώχευσης, τότε σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωτικό να υπάρξει παρέμβαση ρυθμισμένη εκ των προτέρων. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται ένα ισορροπημένο κείμενο. Νομίζω ότι έχουμε και κάποια στοιχεία στην έκθεση για την Τραπεζική Ένωση. Μένουν πολλά να συζητηθούν ακόμα. Ήταν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων, εν πάση περιπτώσει, θα γίνει στις 7 Απριλίου. Έχουμε εδώ ένα χρονοδιάγραμμα. Προβλέπεται επίσης και μια δημόσια ακρόαση στις 23 και 24 Μαΐου. Και 26 Σεπτεμβρίου θα υπάρξει εξέταση της πρότασης και 6 Οκτωβρίου προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Θα μπορούσα να κάνω και εγώ σχόλια για το χρονοδιάγραμμα, αλλά πρέπει να πω ότι η 26 Σεπτεμβρίου και η 6 Οκτωβρίου είναι μεταξύ τους πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση τώρα, αυτό θα το κάνετε κι εσείς. Πάντως τόσες λίγες μέρες ε, νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ ισορροπημένο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται όμως ένα τέτοιο θέμα να το αποφασίσουμε σήμερα. Μπορούμε να κλείσουμε την ανταλλαγή απόψεων επί του συγκεκριμένου θέματος σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε πάλι μια έκθεση του κυρίου Φέρμπερ. Κύριε Φέρμπερ σήμερα μονοπολείται την κατάσταση. Και μάλιστα έχετε δύο εκθέσεις, όχι μόνο μία. Με δύο ξεκινάω, λέει ο κ. Φέμπερ. Όπως γνωρίζετε λοιπόν, έχουμε να συζητήσουμε δύο εκθέσεις σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας MIFID και MIFIR. Δεν χρειάζεται τώρα να κάθομαι να σας εξηγήσω γιατί είμαστε εδώ και τι θα συζητήσουμε. Νομίζω ότι ο εισηγητής θα κάνει την παρουσίαση για τα μύφιλ και μύφιλ με το σωστό τρόπο. Νομίζω ότι κατανοώ τον λόγο για τον οποίο δεν ακολουθείται η απλουστευμένη διαδικασία. Έχει υπάρξει και μια συμπληρωματική τροπολογία. Γι' αυτό θα πρέπει ο κύριος Φέρμπερ να μας δώσει περαιτέρω εξηγήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα του ΜΥΦΙΔ ήθελα να το ξεφορτωθώ από τα τέλη του περασμένου έτους. Αυτό προβλεπόταν, αλλά ούτε μας είχε παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση και αναμένουμε και όλα τα τεχνικά πρότυπα και τα εφαρμοστικά πρότυπα με τα οποία επίσης πρέπει να ασχοληθούμε σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, του ελέγχου. Και πέρσι, στο θέμα του ελέγχου, λάβαμε τον Οκτώβριο μια ειδοποίηση ότι θα υπήρχε καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ΜΥΦΙΤ και του ΜΥΦΙΑ. Και μου προκάλεσε έκπληξη το γεγονό ότι πήρε τέσσερι μήνε μέχρι ότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει αυτό το εκτενές ε, πακέτο. Πολύ λυπάμαι που καθυστέρησαμε τόσο. Θα προσπαθήσω να το περάσουμε λίγο πιο γρήγορα και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σας πω ότι στρώθηκα για να γράψω την, ε, το σχέδιο της έκθεσης. Τα κατάφερα μέσα στην εβδομάδα. Μπορούμε λοιπόν να τα καταφέρουμε πιο δύσκολα, άμα θέλουμε να τα πετύχουμε όλα πιο γρήγορα με όλα τα προβλήματα που έχουμε για το χρονοδιαγράμμα του ΜΥΦΙ και του ΜΥΦΙΑ, πρέπει να πούμε ότι το Κοινοβούλιο ποτέ δεν ήταν το υπήγη των προβλημάτων και τη καθυστέρηση. Ε, ήταν άλλα τα θεσμικά όργανα που καθυστέρησαν. Και θα ήθελα να το έχω πει αυτό εξ αρχής, γιατί με απασχολεί. Όσο για τα θέματα της ουσίας θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Έχουμε πολλά θέματα τα οποία έχουμε διαπραγματευτεί με τις ομάδες. Ανακοινώσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα μπορούσαμε με βαριά την καρδιά να δεχτούμε καθυστέρηση της εφαρμογής κατά νέτος, αλλά μου προκαλεί κάπως έκπλεξη το γεγονός ότι πάλι βγαίνει και λέει η ΕΣΜΑ ότι δεν θα της φτάσει ο ένας χρόνος. Εγώ το είπα ξεκάθαρα και στον Επίτροπο και στον Στίβ ε, Μαγιόρ ότι μία μόνο παράταση θα υπάρξει και να κάτσουν να στρωθούν. Για σε αναβολές ε, πρέπει να σας πω ότι δεν με βρίσκουν σύμφωνο γιατί και θα χαιρόμουν αν η ΕΣΜΑ σε ένα τέτοιο θέμα σιωπούσε και μας έδινε πιο πολλές πληροφορίες επί του περιεχομένου και να σταματούσε να εκφάρει γνώμη για το χρονοδιάγραμμα. Δεν είναι αυτή η δουλειά τη. Η δουλειά τη είναι να μα χορηγήσει τα απαραίτητα στοιχεία. Η πρόταση λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στα πλαίσια των όσων είχαμε συζητήσει και προκαταρτικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, θα πρέπει να σας πω ότι διαπίστωσα ότι υπάρχει και μια ημερομηνία εφαρμογής η οποία προβλέπεται και είμαι πεπισμένος ότι και αυτό θα πρέπει να προσαρμοστεί. Πόσο μάλλον επειδή λείπουν και τα μέτρα επίπεδου 2 που είναι βασικές, ε, βασικοί όροι για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή την ημερομηνία. Άρα και για αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να υπάρξει αναβολή γιατί τα κάτι μέλη δεν μπορούν, δεν μπορούν να τηρήσουν την προθεσμία αυτή, γιατί πολύ απλά δεν έχουν στη διάθεσή τους, δεν έχουν ψηφιστεί τα σχετικά έγγραφα. Και ξέρω επίση ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι που δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια της εφαρμογής διαπιστώσαμε ότι δεν λειτουργεί 100% και μπορεί να γίνει κατευθείαν και μια αναθεώρηση του MIFID αλλά αν διαβάσατε την έκθεσή μου θα δείτε ότι έχω αποστασιοποιηθεί από αυτό. Και αυτό γιατί αν αρχίσουμε να συζητούμε πέρα από τα δεδομένα και άλλα ζητήματα, δεν πρόκειται να ολοκληρώσουμε ποτέ. Και γι' αυτό λοιπόν προτείνω στο σχέδιο του κειμένου να επικεντρωθούμε στο ουσιαστικό που είναι η ημερομηνία. Αν τώρα την ευκαιρία να μιλήσω με την Ολλανδική Προεδρία, θα το κάνω αύριο, γιατί θα με ενδιαφέρε να ξέρω και ποιο είναι το δικό σας χρονοδιάγραμμα. θα ε, ήθελα να έχει το επίπεδο φιλοδοξίας και το Συμβούλιο. Προκειμένου να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Γιατί εγώ ω εισηγητή δεν θέλω από μέρου μου να είμαι καθόλου υπεύθυνο και περαιτέρω καθυστερήσει. Αυτά για τι δύο εκθέσει ε, που υπέβαλα και ελπίζω να είναι οι τελευταίες εκτέσεις για τις οποίες είναι υπεύθυνο για το ΜΥΦΙΤ και το ΜΥΦΙΑ. Να σας υπενθυμίσω ότι από το Σεπτέμβριο του 2011, σχεδόν πέντε χρόνια λοιπόν, θα γιορτάσουμε. Και θα γιορτάσουμε μόνο αν πραγματικά έχουν ολοκληρωθεί τα πράγματα και δεν είμαστε ακόμα εν το μέσο των διαβουλεύσεων. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, εξ ονόματος της Annelies η οποία γέννησε ένα κορετσάκι, αν δεν κάνω σε Συγχαρητήρια. Ναι, ναι, ναι. Μας έστειλε και φωτογραφίε. Όντω, πήρε. Ναι. Η συνάδελφο Αναλή εργάστηκε για το... στο θέμα αυτό και γέννησε την Ισαμπέλα, λοιπόν. Τα πηγαίνουν και δύο μια χαρά. Μάρκο μην ανησυχεί να διαβάσω το σημείωμα της. Το Μύφι 2 και το ΜΥΦΙΑ είναι δύο από τις πιο ευρύες νομοθεσίες μετά την κρίση. Όλες συμφωνούν στο Κοινοβούλιο ότι είναι σημαντικό να τα πετύχουμε σωστά αυτά νομοθετήματα, αλλά ότι και ότι η νέα νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν. Στην Επιτροπή μα πριν από έξι μήνε, ακούσαμε για πρώτη φορά από την ΕΣΜΑ και στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν θεωρούσαν ότι θα κατάφερναν να πετύχουν και να ολοκληρώσουν μέχρι την προσυμφωνημένη προθεσμία τον Ιανουάριο του 2016 μετά από συνάντηση με τους αξιωματούχους της Επιτροπής και της ΕΣΜΑ πρέπει να σας πούμε ότι είχαμε πολλές συναντήσεις μαζί τους και μας προκάλεσε η έκπληξη του γεγονός ότι δεν μας είχαν μιλήσει ποτέ για καθυστέρηση αλλά αποφασίσαμε ότι ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε για να υπάρξει χρηματοπιστωτική σταθερότητα, προστασία των επενδυτών, εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και νομι... νομική βεβαιότητα για τον οικονομικό κλάδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ωστόσο, ήταν σαφέ στην επιστολή του τη 27η Νοεμβρίου του 2015, τον οποίο υποσυπέγραψε ο εισηγητή ε, και ο πρόεδρο, ότι ε, ενώ ήμασταν φυσικά απογοητευμένοι λόγω της καθυστέρησης και μάλιστα λόγω της ε, καθυστερημένης ενημέρωσης για την καθυστέρηση αυτή, γιατί θα δεχόμασταν υπό δύο όρους, ότι η Κομισιόν θα υπέβαλε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τακτικά για την επιτεύξη της πρόοδου και αν χρειάζονταν επιπλέον έτος θα θέλαμε να ξέρουμε τι ακριβώς κόπευε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το έτος και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα ήταν έτοιμα όλα για την ε, νέα η ημερομηνία εφαρμογή. Δεν θα υπάρξει δεύτερη αναβολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα έδωσε ένα αρχικό έγγραφο, αλλά θα χρειαστούμε πολύ πιο πολλέ πληροφορίε κατά την εξέλιξη τη διαδικασία για να είμαστε βέβαιοι ότι θα πετύχουμε αυτά που θέλουμε μέσα στι προσυμφωνημένε ημερομηνίε. Κατά δεύτερον, ξεκαθαρίσαμε ότι σε ό,τι αφορά το ΜΥΦΙΤ και το μυθία θα δεχόμασταν την αναβολή μόνο εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενέκρινε την νομοθεσία επίπεδου 2 όσο το συντομότερο δυνατόν. Και θα απαντούσε στις ανησυχίες του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τις επιστολές, ε, τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στις επιστολές μέχρι την, προς την και προς την ε, Επιτροπή. Δεν έχουν απαντηθεί αυτές οι επιστολές, δεν μας έχει δοθεί διαβεβαίωση ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι ανησυχίε του Κοινοβουλίου και όλου θέλουμε να κινηθούμε το σύντομότερο δυνατόν να δώσουμε νομική βεβαιότητα στους σχετικούς οικονομικούς κλάδους ε, κατά τη φάση εφαρμογής της μεγάλης αυτής της μεταρρύθμισης ε, για να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ευρώπη. Αλλά είναι σημαντικό στο πλαίσιο αυτό να πληρούνται οι δύο όροι που έθεσε η το Κοινοβούλιο. Καλώ ορίζουμε λοιπόν την έκθεση του κυρίου Φέρμπερ καθώ και το πνεύμα συνεργασία, το οποίο επέδειξε ω εισηγητή για το θέμα αυτό. Σε, σε ό,τι αφορά το σχέδιο των εκθέσεων του, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να τροποποιηθεί το κείμενο του ΜΥΦΙΔ 1 για να προσταθούν τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται και να υπάρχει σχετική προσαρμογή. Αυτό το συζητήσαμε και στο παρελθόν και πιστεύουμε ότι γι' αυτό υπάρχει υποστήριξη από όλες τις ομάδες. Θα κάνουμε λοιπόν και μια σχετική τροπολογία προς την κατεύθυνση αυτή. Ελπίζουμε να γίνει δεκτή. Οι βασικές μας ανησυχίες για το MIFID 2 έχουν να κάνουν με το νέο καθεστώς για τα παραγωγά από τον Φιλόν. Ε, και εκφράσαμε τις ανησυχίες μας αυτές σε διάφορες περιστάσεις συμπεριελήφθησαν και σε διάφορες επιστολές εξ ονόματος όλης της διαπραγματευτικής ομάδας προς την ΕΣΜΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέλαμε να μας ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κατά πόσον λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες κατά την κατάρτιση νομοθεσίας δευτερού επίπεδου. Ευχαριστώ και θα τις δώσω τις ευχές σας. Thank you. Thank you, Mr. Η κυρία Σουίνμπον, ευχαριστώ Πρόεδρε και συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή και με τα ε, σχόλια της Αναλύζε που, ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τα 18 κράτη-μέλη ώστε να καθυστερήσουμε τις ημερομηνίε ε, της εφαρμογής της ΜΥΦΙΔ και την εκτέλεσή της. Όσον αφορά την απόφαση το επίπεδο 2, αυτό δεν έχει ακόμα προκύψει από την Κομισιόν και είναι παράλογο να περιμένουμε τα κρατημέλη να εφαρμόσουν τον νόμο χωρίς αυτό. Δεν θεωρώ πως είναι αυτό ε, για να ξαναανοίξουμε την νομοθεσία. Έχουμε περάσει ώρες και ώρες στο τριμερί για να παλεύουμε για τις λεπτομέρειες της μή και όσοι συμμετείχαμε δεν θέλουμε να ξαναρχίσουμε. Κόντεψε να πνιγεί μόνο και μόνο με τις σκέψεις γιατί, οπότε φαντάζομαι ότι συμφωνεί μαζί μου. Ε, είναι λίγοι λοιπόν αυτοί που θέλουν, ε, μάλλον που η νομική ερμηνεία του κειμένου δεν ταυτίζεται με αυτά που είχαμε στόχο. Και αυτά μας άδειξε η ΕΣΜΑ και οι εθνικοί επόπτες και θέλω να υποστηρίξω την ΕΣΜΑ για την αλλαγή επίπεδο 1 που προβλέπει την παράλληλη μεταχείριση των κανονισμό για το... τα, τα πακέτα όπου λαμβάνεται υπόψη οι συναλλαγές ε, πακέτων ε, που είναι ωφέλιμες για τα δεξιωτικά ταμεία ε, δεν αφήσεται αυτό που κάνουν εδώ και δεν θα πρέπει αυτό να μειωθεί όπως ερμηνεύεται στην ερμηνεία του. Κάτι όμως που πρέπει να αναλύσουμε έχει να κάνει με τις εμπορικές εταιρείες υψηλής συχνότητας που φαίνεται ότι έχουν πιάσει διάφορους που προσπαθούν να εμποδίσουν το κίνδυνο, να μειώσουν το κίνδυνο. Οι εταιρείε που τώρα θέλουν να αλλάξουν προϊόντα ξένου συναλλάγματος σε διαφανή ε, με διαφανή τρόπο θα πρέπει να πάνε σε ανοιχτούς ε, εμπόρους ε, over the counter, OTC. Διαφορετικά θα χάσουμε κάθε όφελο των εξαιρέσεων που έχουμε τόσο πολύ σκληρά δουλέψει για να τις εγγυηθούμε. Εάν βρούμε λοιπόν λύσεις σε αυτά τα μικρά ζητήματα που είναι νομικές ερμηνείες θα ήμουν ευγνώμων. Αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι μοναδικές. Δεν ζητώ να ξανανοίξουμε τη συζήτηση περί μύφητα, όμως όταν προκύπτουν τέτοιου είδους προβλήματα νομικής ερμηνείας Νομίζω πρέπει να δείξουμε αρκετή ευθύνη, υπευθυνότητα, ως συνομοθέτες, να έχουμε πολιτική βούληση, ώστε να τα διορθώσουμε. Σας ευχαριστώ. voice again. Well, Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή που κατέθεσε το σχέδιο έκθεσης τόσο γρήγορα μετά τις προτάσεις ε, του, της Κομισιόν. Είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφήνεια για τους εθνικούς νομοθέτες, επόπτες, αλλά και για τους ε, ε, συμμετέχοντες στην αγορά όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής της νομοθεσίας MIFID. Ωστόσο, Εμεί ανησυχούμε για την, ε, την αντιμετώπιση των συναλλαγών πακέτων σε σχέση με τις αλλαγές επίπεδο 1 που θα εισάγουν εξαιρέσεις διαφάνειας για αυτού του είδους τις συναλλαγές. Γι' αυτό και προβλέπ, ε, θέλει να συνεχίσει την συνεργασία με τον συγκεκριτή και τα λαμέλη της διαπραγματευτικής ομάδας για αυτό το ζήτημα στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Φάμπιο Ντεμάζη. Well, even from my side... Και από τη δική μου πλευρά να συγχαρώ την αναλύση και ε, φαντάζομαι ότι γέννησε κανονικά και υποστηρίζω τα όσα ωραία συνόψισε ο εισηγητής Φέρμπερ. Τώρα, τα ζητήματα που αναφέρονται βεβαίως θέλουμε να εφαρμοστούν πλήρως, όπως τα συμφωνήσαμε στο επίπεδο 1 και αυτά είχα να σας πω. Thank you. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε σύντομα λοιπόν να δώσουμε το λόγο στο Τίλμαν Λόιντερ από την Κομισιόν. Μάστε. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτομέρειες. Γιατί μιλήσατε για το δικό μας ε, το χρονοδιάγραμμα και την ταχύτητα με την οποία εκτελούμε την εργασία μας είσαστε, ξέρατε πώς πρέπει να περάσουμε πριν ε, φτάσουμε να υποβάλουμε νομοθετική πρόταση, ίσως να είχατε λίγη περισσότερη κατανόηση απέναντί μας που καθόμαστε εδώ. Ναι, ένας, ε, τέσσερις μήνες μπορεί να είναι πολύ, αλλά είναι πολύ γρήγορα σε σχέση με άλλα κάποιες λεπτομέρειες ότι δεν έχουμε προβεί σε μεγάλες αλλαγές σε αυτή την πρόταση. Γνωρίζουμε το θέμα των συναλλαγών πακέτων, αλλά δεν θελήσαμε να υποβάλουμε πρόταση, γιατί εγώ έχω δει τουλάχιστον πέντε διαφορετικούς ορισμούς για το τι είναι μια συναλλαγή πακέτο. Και για να μπει αυτό σε νομικό κείμενο και να αποφύγουμε να ανοίξουμε το κουτί της Πανδρός είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε προειδοποιώ ότι ο κάθε, η κάθε ένωση ε, κάθε σύλλογος έχει διαφορετική έννοια και ορισμό. Οπότε επίτηδες δεν το προτείναμε. Για το θέμα της επερχόμενης δευτερογενούς νομοθεσίας, οι τρεις κατεξοδότης συμπράξεις είναι σε υποπροετοιμασία, είναι σχεδόν τελειωμένες. Εξετάζουμε τις τελευταίες νομικές λεπτομέρειες και Δυστυχώ υπάρχει μια καθυστέρηση στι μεταφράσει. Πρέπει αυτά να μεταφραστούν στις σε 28 γλώσσε. Οπότε θα μα πάρει άλλο ένα μήνα μήνυμο. RDS. Καταλαβαίνουμε την ανησυχία σας, τη γνωρίζουμε και έχουμε διαβουλευτεί με την ΕΣΜΑ πολλές φορές για τα, την έλλειψη διαφάνειας, ε, για τη διαφάνεια μάλλον στα συναλλαγές μη ε, εκτός χρεογράφων και όλα αυτά θέτουν σε κίνδυνο το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή ότι αυτά όλα θα εφαρμοστούν μέχρι το καλοκαίρι του 2016. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Ε, να πείσουμε την ΕΣΜΑ να μας τα επιστρέψει και να μην έχουμε διαδικασία επίσημης απόρριψης και να καταλήξουμε Ιούνιο-Ιούλιο 2016. Πάντως, για να ξεκινήσει οποιαδήποτε τέτοια επίσημη διαδικασία απόρριψης από την ΕΣΜΑ, δεν θα ανταποκριθούμε στο χρονοδιάγραμμα. Είναι πολύ δύσκολο να επιλύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ξέρω ότι είναι δύσκολο να μας κάνει την πρόταση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν είναι δύσκολο μάλλον να περάσουν όλα αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε πραγματικά ε, την πλήρη κατανόησή μου, αλλά προσπαθούμε και εμείς να περάσουμε διάφορα πράγματα. Από ό,τι κατάλαβα, διάφοροι συνάδελφοι επιθυμούν να συζητήσουμε κάποια θέματα. Το λαμβάνω αυτό υπόψη και για τις συνομιλίες μου με την ε, Ολλανδική Προεδρία, γιατί θα τα πετύχουμε αυτό μόνο αν τα περάσουμε αυτά γρήγορα. Δεν έχει νόημα να κάνουμε επί σειρά μηνών διαπραγματεύσεις. Ούτε η αγορά θα ωφεληθεί από το μήνυμα αυτό, ούτε και εμείς θα ενθαρρυνθούμε. Αλλά το θέμα των συναλλαγών αυτών είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει ακόμα απαντηθεί όπως πρέπει και ξέρω ότι πολλοί το συζητάνε το θέμα του τίτλου, αλλά καταλαβαίνουν κάτι διαφορετικό και θα πρέπει αυτό να το επιλύσουμε, αλλά δεν έχει πολύ νόημα. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να τηρήσουμε το φιλοδοξοφόνο διάγραμμα και ανεξάρτητα από την νομοθεσία αυτή θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα μέτρα επίπεδου 2 τα οποία μας έχει υποσχεθεί να μπορέσει να το τηρήσει. σε ό,τι αφορά τα εφαρμοστικά πρότυπα και τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση με τα οποία θέλουμε να ασχοληθούμε επισταμένως. Αλλά αυτό είναι ξεχωριστό κεφάλαιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν συνάδελφοι για τις παρεμβάσεις. Μου καταδεικνύουν ότι οι πολλές ώρες που συζητήσαμε έχουν αποφέρει καρπούς και θα είμαστε σε επαφή τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Thank you. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν τη συνεδρίαση γιατί, ή μάλλον την συζήτηση για τη συγκεκριμένη έκθεση. Η διαδικασία από εδώ και πέρα θα γίνει για τη συγκεκριμένη έκθεση μόνο στην αγγλική γλώσσα τροπολογίες ε, δεν μπορούν να κατατεθούν ε, ηλεκτρονικά αλλά μόνο ε, σε γραπτό κείμενο προς τη γραμματεία. Προθεσμία είναι 29 Φεβρουαρίου, 5η απογευματινή. Εξέταση των τροπολογιών 16 και 17 Μαρτίου. Η ψηφοφορία θα γίνει στην Ολομέλεια σε χρόνο που θα αναφερθεί αργότερα τέλος της συνεδρίασης, η επόμενη συνάντησή μας προβλέπεται για τη 15η και 16η Μαρτίου.